Καλησπέρα σε όλους. Χαίρετο και τον κύριο Λαμασούρα από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Όπως ξέρετε είναι μια κοινή συνεδρία της Επιτροπής Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Και πριν ξεκινήσουμε τις ψηφοφορίες, ήθελα να δώσω τον λόγο σε δύο, στους δύο συγητές, την κυρία Γκρέσλε και τον κύριο Ριβελίνη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Απλώς ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι με βοήθησαν στο δύσκολο έργο της προετοιμασίας της ψηφοφορίας τους υπαλλήλους της Γραμματείας και ιδίω επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γκρέσλε η οποία πραγματικά έπαιξε ένα ουσιαστικό ρόλο στην περάτωση αυτής της εργασίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο εισηγητές. Ε, κύριε Γκάιερ. Πράγματι όλοι οι προαναφερθέντες αξίζουν ευχαριστήσεις, αλλά υπάρχει μια διόρθωση. Η τροπολογία υπαριθμών 56, η δική μου είναι σελίδα 3 κάτω-κάτω, έχει αποσυρθεί. κατάφερε να απαλύνει τις αμφιβολίες μου εισηγητής, οπότε αποσύρω την τροπολογία υπαριθμών 56. Ευχαριστώ κύριε Γκάιερ. Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, είναι κυρία Γκρέσλερ. Στο εκτιμώντας ένα υπάρχει μια τροπολογία 1 του εισηγητού την οποία επίσης αποσύρουμε και ανταυτού θέλουμε να υιοθετηθεί η τροπολογία 1 της ΑΦΕΤ γιατί είναι πιο ακριβής. Ευχαριστώ. Eh, io vado a chiedere, non è, non è chiaro. Amendment 1 ist das Recital. Η τροπολογία 1 στο εκτιμώντα 1 να αντικατασταθεί από αυτήν τη ΑΦΕΤ τη Επιτροπή Εξωτερικών. Η σελίδα 6 είναι η τροπολογία. Ωραία, καλώ. Ναι, Κύριε Κουλτιέρη, να σας πω και μόνο ότι μετά από την απόσυρση της τροπολογίας 56 από τον κύριο Γκάιερ, η ομάδα μας μπορεί να υποστηρίξει την τροπολογία 21. Στη σελίδα 3 η τροπολογία 56, την απέστειλε ο κύριος Γκάιερ, την 56, ως εκ τούτου εμείς θα ψηφίσουμε την 21 των εισηγητών. Ωραία λέει ο πρόεδρος. Εντάξει, αν έχουν τελειώσει παρεμβάσει τελευταία στιγμή, μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Λοιπόν, ξεκινάμε με την ψηφοφορία με την τροπολογία 10, όπου έχουμε μια προφορική τροποποίηση. Άρχεται η ψηφοφορία. Cosa stiamo facendo? La votazione è chiusa. Πέρας ψηφοφορίας. Approvato 41. Εγκρίνεται 41 με 9 με μία αποχή. 11 απεσύρθη. Η τροπολογία 12. Τώρα τον εισηγητών άρχεται η ψηφοφορεί. La votazione è chiusa. Πέρα τη ίδια αυτή τη ψηφοφορία. Approvato con 53 voti. 53-1 εγκρίνεται. Παρακαλώ. Ήθελα να σας πω μονάχα. Ήθελα να πω. Πως ε, δεν ε, είναι εδώ πέρα η τροπολογία μου. Είναι κατά κανόνα πάνε... Έχω την κάρτα μου εδώ πέρα, κατά κανόνα την έχω μαζί μου, αυτή τη φορά όχι. Τροπολογία 13. Δεν έχω φέρει Allora, la votazione aperta. Άρχεται η ψηφοφορία, όχι, πέρασε η ψηφοφορία. Εφόσον δεν έχει εγκριθεί η προφορική τροπολογία 1, εκπίπτει, λέει η κυρία Γκρέσλε. Ρέγω. Συνεχίζουμε με τη συμβαστική 1, λέει η κυρία Γκρέσλε. Σε λέω non c'è questo. No, but, uh... L'emendamento 13, no? L'emendamento 13. Εφόσον δεν εγκρίθη η προφορική τροπολογία 1, εκπίπτει η 13, λέει ο πρόεδρο. Εάν δεν εγκριθεί η τροπολογία 1, η προφορική τότε εκπίπτει. Μα εγκρίθηκε, λέει ο κ. Λαμασούρ. Ε, λέει ότι εκπίπτει εάν δεν έχει εγκριθεί. Λοιπόν, μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα. Εγώ ελπίζω να μην χρειαστεί ποτέ να αντιμετωπίσω ένα τόσο πολύπλοκο φάκελο, λέει η κυρία Γκρέσλε. Ναι, ναι, είναι μπερδεμένα. Λοιπόν, 13 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 51 υπέρ, 8 κατά εγκρίνεται. Προχωρούμε στην τροπολογία 50, άρχεται η ψηφοφορία.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 Πέρας. Εγκρίνεται με 55 ψήφους υπέρ και 2 ψήφους κατά. Τροπολογία 14 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 51 ψήφι υπέρ, 9 κατά. 53 ψήφι υπέρ. Άρχεται ψηφοφορία μάλλον. Πέρας. Εγκρίνεται με 31 ψήφους υπέρ, 29 κατά. Λοιπόν, eh, καταπίπτει η επόμενη τροπολογία γιατί η 53 έγινε δεκτή. Οπότε περνάμε συμβαστική 2 και στην 7 άρχεται ψηφοφορία. La votazione Πέρας. 57 υπέρ 1 κατά 2 αποχές. Περνάμε λοιπόν τώρα στην προφορική τροπολογία 3 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 59 υπέρ 2 κατά. Δεύτερο τμήμα, ψήφι υπέρ. Μάλλον άρχεται η ψηφοφορία. La votazione chiusa. Πέρας. Ψηφίζει ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Εντάξει. Πέρας ψηφοφορίας. 31 ψήφοι υπέρ, 30 κατά. Ε, κάτε questo. 55 ε, Η 55 εκπίπτει. La votazione è aperta. Επιτροπή Ανάπτυξη. Άρχεται η ψηφοφορία. Παρακαλώ. Το τρίτο τμήμα τη χωριστή ψηφοφορία τι το κάναμε. Α, έχει αποσυρθεί, συγγνώμη. Είναι μπερδεμένα, κύριε Πέρα για την ε, Επιτροπή Ανάπτυξη. Ε, Απορρίπτεται με δύο ψήφους υπέρ 57 κατά. Τροπολογία 20 με ε, τροποποίηση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Mm. 59 υπέρ 2 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 12 Al 21, mi dicono che è caduto. Quindi emendamento 21. Ναι, 20 εξέπεσε. Τροπολογία 21 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 52 υπέρ 9 κατά. 56 έχει αποσυρθεί. Συμβιβαστική τροπολογία υπαριθμών 3 η σοσιαλιστική ομάδα ζήτησε ψηφοφορία σε τρία χωριστά τμήματα. Πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 58 υπέρ μία ψήφος κατά μία απόχη. Mm. Δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. La Πέρας. Από το ΕΚ ψηφίζει ένα άτομο παραπάνω. Λοιπόν, 34 υπέρ, 25 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα τώρα, άρχεται την ψηφοφορία. La Πέρας. Εγκρίνεται 31 υπέρ, 29 κατά και μία αποχή. L'emendamento 23 soppresso, Τροπολογία 23. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρα. Πέρας. 36 υπέρ, 24 κατά, μία αποχή εγκρίνεται. 24. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρα. Πέρας. Εγκρίνεται. 58. Άρχεται η ψηφοφορία. Εκπίπτει 58 λέει η κυρία Γκρέσλη. Εκπίπτει λέει η κυρία Γκρέσλε. Συμβιβαστική τροπολογία 4. Και εδώ έχουμε δύο χωριστά τμήματα. Πρώτο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Πέρας. Εγκρίνεται. 59 υπέρ. Δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Votazione Πέρας απορρίπτεται 30 υπέρ, 31 κατά και μία αποχή. Adesso 26. 26. 26, Τροπολογία 26. Άρχεται ψηφοφορία. Παρακαλώ. Πόσοι ψηφίσανε από το ΕΛΚ στο δεύτερο τμήμα της συμβαστικής τροπολογίας 4. Ja, ist without card. Okay. Es war eines der Schlüsselamendments deswegen. Γιατί είναι μια κομβική τροπολογία. Okay. Okay. Andiamo avanti, dai. Emendamento 26. Come no? Al microfono. Sì, sì, come no. Giustamente Ακριβώς. Προσπαθώ να καταλάβω αν ψήφισαν όλοι από το ΕΛΚ όταν είπατε ότι ήταν ένας ο οποίος ψήφιζε παραπάνω έφυγε ο συνάδελφός μας. Μήπως υπήρξε κάποιο σφάλμα, μήπως ε, ξέχασε να μην ψηφίσει. Πάση έχει κλείσει αυτή η ψηφοφορία. Εκτός αν υπάρξει κάποιος ο οποίος ξέχασε να ψηφίσει και τότε είναι διαφορετικά τα πράγματα. Σας είπα και πριν κύριε Πρόεδρε ότι δεν έχω την κάρτα μου αλλά είμαι παρόν στην αίθουσα και είπα μου είπατε ότι έπρεπε να φύγει ένας από το ΕΛΚ έφυγε πάντα σήκωνα το χέρι μου σε όλες τις ψηφοφορίες ε, ήταν φανερό το πως ψήφιζα Γι' αυτό ήταν δικαιολογημένο το ερώτημα της κυρίας Γκρέσλε. Προτείνω να επαναλάβουμε αυτή την ψηφοφορία. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι ένα πρόβλημα. Όταν εσείς σηκώνετε το χέρι σας, αυτό δεν ε, καταδεικνύεται στον υπολογιστή αν είναι περισσότερα τα μέλη του ΕΛΚ ή λιγότερα τα οποία ψηφίζουμε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Θα πρέπει συγχρόνω σε κάθε ψηφοφορία να ελέγχουμε πόσοι ψήφισαν από την πολιτική σα ομάδα. Καταλαβαίνετε. Αλλά ακόμα και αν υπήρχε μια ψήφο παραπάνω από το ΕΛΚ, σε ισοψηφία πάλι θα, δεν θα περνούσε αυτή η τροπολογία. Δεν έχει εγκριθεί, εν πάση περιπτώσει. Χρειαζόταν δύο ψήφοι ακόμα για να περάσει. Δεν φτάνει μία χωρίς μικρόφωνο μιλτής. Αν θέλετε να επαναλάβετε την ψηφοφορία νομίζω είναι καλύτερο. Όχι. Αυτό έχει τελειώσει η ψηφοφορία. Ε, προχωρούμε. Επόμενη τροπολογία, αρχή ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται με 35 ψήφους υπέρ 26 κατά. Εκπίπτει ως εκ τούτου η, τροπολογία, η επόμενη τροπολογία 60 τώρα. Άρχεται την ψηφοφορία. La votazione è chiusa. Πέρας. Απόλυτα. 26 υπέρ 36 κατά. Επιτροπή Ανάπτυξης 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται 40 ψήφοι κατά, 18 υπέρ. 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 37 ψήφοι υπέρ, 24 κατά. 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 55 ψήφοι υπέρ. 61. Άρχεται η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 30, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 36 ψήφους υπέρ. Διολογικές σκέψεις, τροπολογία 31, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με 58 αρνητικέ ψήφου. Τροπολογία 1 τη επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1 έχει αποσυρθεί των εισηγητών. εκπίπτει και 32. Πάμε στην συμβαστική τροπολογία 5 για την αιτιολογική σκέψη 2. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Όχι, όχι, καλύπτεται, καλύπτεται από τη συμβαστική. Συμβαστική τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 7. Άρχεται ψηφοφορία. Α, την έχουμε ήδη ψηφίσει, ναι. Συμβαστική 8. 8. Άρχεται ψηφοφορία. Συμβαστική 8. Πέρας. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική παριθμόν 9, άρχεται ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39, άρχιδη ψηφοφορία. λήξει. Ένας παραπάνω ψηφίζει από το και πάλι. Θα πρέπει να εξαλειφθεί αυτός ο συνάδελφος. Απορρίπτεται, εν πάση περιπτώσει. Τροπολογία 40. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 41. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 32-30. Τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 43. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 44. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 45. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 46. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλειος η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Εξωτερικές ε, συνταγματικές υποθέσεις 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απέριπτε. Συμβιβαστική 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6 της Συνταγματικής Επιτροπής. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 48 εκπίπτει και 6. 9. Ψηφοφορία άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 49. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 59 ψήφους υπέρ, 3 κατά και καμία αποχή. Τελικό ψήφισμα λοιπόν. Το ψήφισμα όπως έχει τροποποιηθεί. Πέρας. εγκρίνεται με 53 ψήφους υπέρ, 3 ψήφους κατά. Κύριε Πρόεδρε μου, ευχαριστώ, συγχαίρω τον εισηγητή και μπορούμε νομίζω να συμπεράνουμε ότι οι εισηγητές πρέπει να συνεννοηθούν τώρα με την Κομισιόν και το Συμβούλιο για να επιζητήσουν επί της βάσης αυτής μια συμφωνία που να επιτρέπει ενιαία ανάγνωση και για τα δύο όργανα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Se prendiamo posto, continuiamo la riunione della Commissione. Καθίστε να συνεχίσουμε παρακαλώ. Υπάρχουν θέσεις πίσω. να σας πληροφορήσω συμπαθάτε με αλλά να λίγη ησυχία σ, σ, σ. Allora, vi devo informare delle... Πρέπει να σας πληροφορήσω για τις αποφάσεις των συντονιστών στο Στρασβούργο 3η 7 Σεπτεμβρίου αποφάσεις για τις διαδικασίες ορισμού εισηγητών. Η δική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου Βόγκαν για τους σοσιαλδημοκράτας, Deutsch για την ειδική έκθεση διαρροτικών μετρών Ευρωπαϊκή Ένωση, και τις δαπάνες για την προμήθεια νερού, Κάλβιν, σοσιαλδημοκράτες, κυρία Κέστινγκερ του ΕΛΚ για άλλη ειδική έκθεση του ελεγκτικού. Για την προστασία δε των συμφερόντων της Ένωσης και την καταπολέμηση της απάτησης συντονιστές ενέκριναν έκθεση πρωτοβουλίας το, ήδη από το 9 και αυτά όλα βέβαια θα εξαρτηθούν από την αυτόματη έγκριση της Προεδρίας και των Προέδρων των Επιτροπών, αλλά ακόμα δεν την έχουμε λάβει. Κύριε Πρόεδρε, για αυτό το οποίο μόλις είπατε στη συνεδρίαση των συντονιστών, συζητήσαμε και το πώς θα κυλήσει χρονικά η απαλλαγή του προπολογισμού του 2009 η κυρία Γκρέσλε είπε πως ο, κύριος, ο Επίτροπος Άντε ε, για τα κοινωνικά και ο Τσόλος για τα αγροτικά και υπάρχει και βεβαίως ο Επίτροπος ε, για τα εξωτερικά και συνιστώ τον κύριο Πίμπαλξη για την ε, ανάπτυξη το λέω απλά για να γραφτεί στα πρακτικά, γιατί είναι τομέα ε, που αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και προτείνω όλα αυτά να μπουν στον Δεκέμβριο. Ελπίζω να συμφωνεί η κυρία Γκρέσλε. Παρακαλώ κυρία Γκρέσλε. Ήθελα να υπενθυμίσω πως ε, μόλις ε, ψηφίσαμε για να μπει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στον προϋπολογισμό, οπότε νομίζω το έχουμε φροντίσει. Καλώς, συμφωνούμε όλοι. Καρνισόρη Ιβαν. Ε, έχουν οριστεί για αυτή την ε, έκθεση για την δε έκθεση είναι για την απαλλαγή 2009 εκεί πέρα έχουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες για την απαλλαγή 2009 οι συντονιστές επιπλέον ε, ενέκριναν την έκθεση του ΕΛΚ για μια έκθεση πρωτοβουλίας για τους ε, τομείς ε, της καταπολέμησης ε, της απάτης και αποφάσισαν οι συντονιστές να μην υπάρξει σύνταξη γνωμοδότησης αλλά ένα για το έγγραφο της Κομισιόν για τη μεταρρύθμιση του Όλαφ αλλά να απευθυνθεί μια επιστολή στον πρόεδρο Μπούζεκ έτσι ώστε ο Επίτροπος να πληροφορηθεί σχετικά. Κατόπιν έχουμε αντιπροσωπείες και ακροάσεις για το 2011 οι οποίες επίσης αποφασίστηκαν τέλος Οκτωβρίου Ιταλία μετά πρόγραμμα για τους μπλοκαρισμένους νομοθετικούς φακέλους στο Συμβούλιο μετά έχουμε την απαλλαγή όπου η Κομισιόν για το 2009 πρότεινε να γίνει μια συζήτηση για την ανακοίνωση της Κομισιόν για την ισορροπία των ελέγχων και ειδικά όσον αφορά τη συχνότητα των περιπτώσεων και μετά έχουμε την διαδικασία ορισμού του νέου διευθυντού τις όλα οι σοσιαλιστές ενέκριναν το αίτημα των σοσιαλιστών να ζητήσουμε από το ελεγκτικό συνέδριο να συντάξει μια ειδική έκθεση για την χρήση των κονδυλίων για την προστασία από τις καταστροφές και συμφώνησαν να υπάρξει μια συνεδρίαση με τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου για να συζητήσουμε για την κατάσταση η οποία επικρατεί ακριβώς για το θέμα της απαλλαγής. Oh. Κατόπιν περνάμε σημερινή συνεδρίαση. Την συνεδρίαση που έλαβε χώρα σήμερα το πρωί. Εκεί πέρα μιλήσαμε για τις ακροάσεις και για τα ταξίδια των αντιπροσωπιών για το 2011. Έχουμε τρία ταξίδια αντιπροσωπιών για το 2011 Ξεκινάμε τον Απρίλιο Ουγγαρία, Κοσφοπέδιο, Πουγούδουμου και Γαλλία ναι, και αρχές 2012. Ε, Για το 2011 οι ακροάσεις θα είναι τέσσερις. Μεταρρύθμιση του ελεγκτικού συνεδρίου και σχέση με τα θεσμικά όργανα, βελτίωση του μηχανισμού συμπερίληψης, μετά ακρόαση για τα αποτελέσματα της διαδικασίας απαλλαγής 2008 για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες, μετά ακρόαση για την αποτελεσματικότητα των ε, ταμείων, ειδικά στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ε, μία επίσης για το καθεστώς των υπαλλήλων και άλλη μία για το θέμα των whistleblowers. Μετά έχουμε την διαδικασία ακρόασης υποψηφίων για την θέση διευθυντού της Όλαφ. Υπόθηκε πως πρέπει να διατηρήσουμε την ίδια διαδικασία του 2005 μετά την σημερινές ε, ψηφοφορίες ζητήθηκε από τους ε, συναδέλφους ε, Ριβελίνη και Γκρέσλε να εξετάσουν τις προτινόμενες αλλαγές με στόχο να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε στην πρώτη ανάγνωση. Μετά έχουμε την απαλλαγή 2009 για το χρονοδιάγραμμα αποδεχτήκαμε τα όσα είπε η εισηγητής Ήταλα, ο δε γενικός γραμματέας στις 25 και 26 Οκτωβρίου θα πρέπει να είναι παρόν συνεδρίαση των συντονιστών και θα προσκληθεί και στην συνεδρίαση της 30 Ιανουαρίου 2011 για το Αφγανιστάν εκεί πέρα ξεπεράσαμε τη σύγκρουση με την Επιτροπή Εξωτερικών. Οι συντονιστές αποφάσισαν η Επιτροπή Ανάπτυξης να υποβάλει έκθεση. Επίσης έχουμε επίσκεψη στην Ιταλία από τις 26 μέχρι 28 Οκτωβρίου, η οποία είναι αποδεκτή. Και υπάρχει επίσης ένα γραφείο ερευνητική δημοσιογραφίας, το οποίο θα το συναντήσουμε σε εξωτερικές δραστηριότητες επίσκεψη στην Ιταλία μετά για τον Όλαφ είχαμε πει πως αναμένουμε βεβαίως την νομοθετική διαδικασία και εκεί πέρα έχει υποβάλει την πρότασή του το Κοινοβούλιο για την πρώτη ανάγνωση μετά Ανακοινώθηκε πως ο κύριος Μπάλφορ θα είναι παρόν στην επόμενη συνεδρίασή μας ως ε, πρόεδρος του Συμβουλίου. Οπότε φτάνουμε στο σημείο 22 της ημερήσιας διάταξης, ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελληνικού Συνεδρίου υπαριθμών 15-2010 με θέμα βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιούμενη μέσω οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών λήψη αποφάσεων και παρακολούθηση. Η κυρία Γκρέσλε έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πίνξτεν και το ελεγκτικό συνέδριο αλλά και την γραμματεία της Επιτροπής μας. Έχουμε συνεργαστεί βεβαίως και με τον τότε πρόεδρο της Επιτροπής ε, που είχαμε μία μήνυ αντιπροσωπεία και είχαμε πάει και στη Νέα Υόρκη με την Κομισιόν για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα με τον ΟΗΕ. Προσπάθησα λοιπόν να αναφέρω κάποια από τα αποτελέσματα του ταξιδιού και της έκθεσης της Κομισιόν, του ε, με ελεγκτικού συνεδρίου γιατί αυτό το οποίο ε, είχαμε πάντα ως αίσθηση, το επιβεβαίωσε το ελεγκτικό συνέδριο, δηλαδή πως έπρεπε να ρίξουμε μια ματιά στη χρήση του ταμείου και βλέπουμε πως δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι γίνεται με τα λεφτά μας. Εντάξει, υπάρχουν γυαλιστερά προσπέκτους από τις διάφορες υπηρεσίες του ΟΗΕ, αλλά το πώς μας δίνουν λόγο και το τι κάνει η Κομισιόν έναν των κρατών μελών για τα ευρωπαϊκά χρήματα δεν είναι μια προσέγγιση ανάλογη με την δική μας αυτή η οποία ακολουθείται στον ΟΗΕ. Οπότε περιορίστηκα στα βασικά. Καθώς υπάρχει και αυτή η τριετής ε, αξιολόγηση. Οπότε θα πρέπει να υπάρχουν σαφές ε, σαφείς ε, γραμμέ για τα καταπιστεύματα αυτά πολλαπλών δωρητών. Η Κομισιόν έχει ήδη αυτή τη δυνατότητα ελέγχου, αλλά δεν την χρησιμοποιεί. Οπότε αυτό το οποίο σκεφτόμαστε είναι π.χ. στο κοσφοπέδιο που είναι και στην πόρτα μας και είναι, είμαστε και οι μεγαλύτεροι δωρητές ε, να δούμε τι γίνεται να μπορούμε να το λειτουργήσουμε με απλοποιημένους κανόνες γιατί οι κανόνες αυτή τη στιγμή είναι πολύ πολύπλοκοι επίσης Δυστυχώς το δικαστήριο δεν τα συμπεριέλαβε αυτά στις ε, δικές του συστάσεις, γι' αυτό θέλω να αναφερθώ ακριβώς στο ελεκτικό συνέδριο και να ε, μάθω και ποιες είναι οι δικές τους εμπειρίες. Επίσης θεωρούμε πως χωρίς σαφή πρόοδο στη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ θα πρέπει να σκεφτούμε αν θέλουμε να συνεχίσουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή βλέπουμε το πώς χρησιμοποιούν τα λεφτά μας και το τι λογαριασμό δίνουν ήταν κάτι το σοκαριστικό. Θα αναφέρω και παράδειγμα στο οποίο αναφέρθηκα το κοσφοπέδιο. Έγινε μια αποστολή Ε, υπό τον τίτλο ITF ε, μία δηλαδή αποστολή της ε, Guarda di Finanza του Όλαφ και του εσωτερικού ελεγκτή του ΟΗΕ για τη χρήση των κονδυλίων για το κοσφοπέδιο. Ε, εμφανίστηκαν λοιπόν διάφορες μεμονωμένες εκθέσεις τις οποίες μπορείτε να τις δείτε στο Wikileaks εάν τις θέλετε αν θέλετε τα links τα έχω εγώ Μπορείτε να δείτε λοιπόν τι υπάρχει σε αυτές τις εκθέσεις και αν δείτε το τι έκαναν τα κράτη-μέλη μας στην έκθεση ελέγχου του προβλησμού του ΙΕ είναι σκάνδαλος. Έλαβαν υπόψη τους δηλαδή τις εκθέσεις, έτσι είπαν, και είπαν πως ε, ε, είχαμε απάτες έτσι, σε οποίες συμμετείχε το προσωπικό του ΙΕ και δεν δόθηκε καμία συνέχεια. Μιλάμε για σοβαρές περιπτώσεις απάτες και ε, πράγματα όπως σεξουαλική παρενόχληση γυναικών υπαλλήλων και μιλάμε για μουσουλμανική χώρα ε, το κοσφοπέδιο. Αν ακούμε δηλαδή ότι το προσωπικό του ΟΗΕ ε, το προσωπικό του ΟΗΕ δηλαδή να φτάσει να εκβιάζει σεξουαλικές σχέσεις με αντάλλαγμα μία δουλειά και αυτοί οι άνθρωποι υποτίθεται ότι διαφυλάτουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και πάει αυτό στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΗΕ και δεν κάνουν τίποτα, απλά το, το λαμβάνουν υπόψη. Ε, πρέπει να κινητοποιηθούμε. Λοιπόν, υπάρχουν αυτά τα έγγραφα, εμφανίστηκαν και στη Νέα Υόρκη και ποτέ δεν υπέφτα πως θα είναι τόσο ψυχρή και δεν θα κάνουν τίποτα. Και μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα παρά το ότι τακτικά προσπαθούμε να το κάνουμε θέμα αυτό και σήμερα. Νομίζω και ο κύριος Χατζημαρκάκης εδώ πέρα και ο κύριος Λάμστορφ ε, τα, τα ξέρουν αυτά. Κάθε φορά ε, βλέπω εδώ πέρα έτσι, κάθε φορά που τα αναφέρω αυτά τα θέματα, πρόσωπα, έτσι χωρίς κατανόηση. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρξει μια εσωτερική μεταρρύθμιση του ΟΗΕ και να δούμε βεβαίω και το τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς από την πλευρά μας για την κατανόηση και τη διάδοση αυτού του ζητήματος. Και το έχω συζητήσει και με τον Γενικό Διευθυντή και με τους συντονιστές σήμερα το πρωί και όταν ακούω πως ε, επετράπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παραστεί ως παρατηρητή στην ε, ε, Γενική Συνέλευση και βλέπω πως καταψηφιστήκαμε 61 έναντι 76 ειδικά από τις χώρες ακές τις οποίες στέλνουμε τα λεφτά πλέον δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Οπότε το θέμα αυτού του ταμείου του ΟΗΕ είναι σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ξέρω πως υπάρχουν πλέον περιοχές ε, εντάξει, που ε, ε, που είναι ευγνώμονε στον ΟΗΕ που υπάρχει εκεί πέρα και δραστηριοποιείται και δίνει λεφτά όπω παραδείγματο χάρη η Παλαιστίνη. Οπότε θα πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση με τον ΟΗΕ, να δούμε αν έχει υπάρξει κάποια ουσιαστική πρόοδο να δούμε και έγγραφα. Ε, ούτε καν η Κομισιόν δεν έχει αυτό το δικαίωμα να δει έγγραφα του ΟΗΕ, να γνωρίζουμε τι κάνουν τα λεφτά μα. Είδαμε την έκθεση βεβαίως ε, δραστηριοτήτων 2009 με την συνήθεια επιφύλαξη, τα ξέρουμε αυτά. Αναμένω κάποιες ε, εξηγήσεις, δεν υπάρχουν ε, ούτε και σήμερα βεβαίως πάλι τα ίδια. Θα πρέπει να το συζητήσουμε λοιπόν κάποια στιγμή σοβαρά, οπότε άκουσα και θα ήθελα να ακούσω και από την Κομισιόν και το Ελεκτικό Συνέδριο ποιες αλλαγές θέλουν για να μπορέσουν επιτέλους να δώσουν ε, λογαριασμό το τι κάνουν τα λεφτά μου. Αυτά σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, ναι. Το Ελεκτικό Συνέδριο. Πριν ε, δώσω τον λόγο στον κύριο Κάιρ, βλέπω τον κύριο Κάλλη Πίνξεν από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου καταρχάς ε, να επωφεληθώ για να συγχαρώ την εισηγήτριά σας κυρία Γκρέσλε γιατί με μεγάλο ενδιαφέρον και εγώ και η ομάδα μου διαβάσαμε το έγγραφο εργασίας της το οποίο συνοψίζει κάλλιστα τα συμπεράσματα του ελεγκτικού συνεδρίου από τον δημοσιονομικό έλεγχο που έκανε για τα ταμεία που, για τους, τα ποσά που διαθέτουμε στον ΟΗΕ ή για τα ταμεία που διαχειρίζεται ο ΟΗΕ. Η κυρία Γκρέσλε λοιπόν νομίζω ότι έκανε τη δουλειά της όπως ακριβώς ήρμαζε σε μια ευρωβουλευτίδα. Πρέπει όμως να σας πω επίσης ότι κατανοώ πολύ καλά και τις επικρίσεις της ως προς τον ΟΗΕ. Δεν ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί, αλλά όπως εσείς και πριν από εσάς ίσως, πήγαμε και εμείς στη Νέα Υόρκη, εγώ και ο διευθυντής τότε του γραφείου μου και τώρα υπεύθυνο για εξωτερικές δράσεις, ο κ. Φραντίου και ως ελεγκτικό συνέδριο εμείς ε, πρέπει να εκφραζόμαστε πάντοτε με πολύ φρόνιμο τρόπο και θα έλεγα λοιπόν ότι κατά την επίσκεψη αυτή νιώσαμε κάτι ανάλογο με αυτά που νιώσατε κι εσείς ως ευρωβουλευτέ. Καταλαβαίνω λοιπόν πολύ καλά τι εννοούσατε. Και τώρα αν επιτρέπετε κύριε Πρόεδρε θα ήθελα συντομότατα να σας κάνω μια εισαγωγή στο έγγραφο του συνεδρίου. Λέω σύντομα γιατί τα έχει πει όλα η κυρία Γκρέσλε και φαντάζομαι ότι όλοι οι βουλευτές εδώ και βουλεύτριες θα έχουν διαβάσει το έγγραφό μας και το έγγραφο εργασίας της κυρίας Γκρέσλε. Επιτρέψτε μου λοιπόν να είμαι συντομότατος. Πρώτα πρώτα πριν γίνει η σύντομη εισαγωγή, πρέπει να σας πω ότι το έγγραφο αυτό είναι το πρώτο τμήμα του ελέγχου όπου έπρεπε να απαντήσουμε σε δύο συγκεκριμένα ερωτήματα. Θα σας τα πω σε λίγο. Τώρα τελειώνει η δεύτερη, το δεύτερο τμήμα, ο δεύτερος έλεγχος Έγινε μια πρώτη συζήτηση βέβαια την περασμένη εβδομάδα. Θα συνεχιστεί και η δεύτερη αυτή λοιπόν έκθεση θα αφορά γενικότερα ε, θα τελειώσει μάλλον μέσα σε δύο-τρεις μήνες περίπου, περίπου, περίπου. Στο έγγραφό σας κυρία Γκρέσλε αναφέρεται και το κοτσιφοπέδιο, ο έλεγχος όμως που έγινε δεν αναφέρει ούτε μια λέξη για αυτή την περιοχή αλλά θα μπορούσα να σας πω για να το μάθουν και οι αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ ότι κάθε χρόνο κάθε χρόνο εξετάζουμε σύντομα το θέμα του επόμενου χρόνου και αυτή τη φορά ήταν το κοσυφοπέδιο. Θα γίνει λοιπόν ένας δημοσιονομικός έλεγχος που θα αφορά και το κοσυφοπέδιο διότι ξέρουμε ότι ξέραμε ότι το κοινοβούλιο ενδιαφερόταν. Τώρα ο δημοσιονομικός κανονισμός ακόμη τον συζητάμε. Δεν μπορώ λοιπόν να σας σχολιάσω τίποτα ακόμα τον συζητάμε όμως ακόμα. Και τώρα έρχομαι χωρίς άλλη καθυστέρηση στον ίδιο τον δημοσιονομικό έλεγχο. Δύο ερωτήματα όπως σας είχα πει είχαμε θέσει. Πρώτον, όταν η Κομισιόν αποφασίσει να συνεργαστεί με τον ΟΗΕ έχει προηγουμένως χρησιμοποιήσει κανένα συγκεκριμένο κριτήριο έχει σκεφτεί ποια θα ήταν τα ωφέλη και τα μη ωφέλη από τέτοια συνεργασία. Δηλαδή ταχύτητα, ποιότητα, παρουσία, επιτόπου κλπ. Προφανώς αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν συνεργάζεται με τον ΟΗΕ, είναι προφανές θα υπάρχουν και ωφέλη και όχι. Και το θέμα που θέσαμε ήταν, ήταν λέγω, αυτή τη συνεργασία την πραγματοποιεί η Κομισιόν, όχι. Άρα τα ωφέλη από συνεργασία με τον ΟΗΕ ε, δεν είναι προφανή. Ενώ θα έπρεπε, θα έπρεπε. Για λόγους και νομικούς και στρατηγικούς. Δεύτερο ερώτημα που θέσαμε στον εαυτό μας. Euh, το monitoring, monitoring που λέμε. Αυτό το monitoring λοιπόν μας δίνει επαρκείς πληροφορίες για να γνωρίζουμε αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι και για να γνωρίζουμε ποιες είναι οι δημοσιονομικές ή χρηματικές διαδικασίες. Και εδώ η απάντηση είναι αρνητική. Ας πω λοιπόν σε άλλη γλώσσα τώρα για το πρώτο ερώτημα ότι το συνέδριο κατέληξε ότι η Κομισιόν δεν χρησιμοποιεί, για να το πω έτσι απλά, κανένα πρακτικό κριτήριο κατά τη λήψη των, της απόφασης αν θα συνεργαστεί ή όχι με τον ΟΗΕ. Είναι λοιπόν σαφές από την έκθεσή μας ότι το ότι η Κομισιόν δεν προβαίνει πριν αποφασίσει να συνεργαστεί με τον ΟΗΕ ή με οποιαδήποτε άλλη οργάνωση γιατί αναφέρουμε περίπου 30 εδώ στην εκκλησία μας, δεν προβαίνει σε μία ανάλυση που να δείχνει ποια είναι τα ωφέλη. Αυτό σημαίνει ότι η επιλογή μία οργάνωση του ΟΗΕ δεν βασίζεται σε επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η συνεργασία είναι πιο αποτελεσματική από οποιαδήποτε άλλη συνεργασία. Άρα, όπως είπε και η κυρία Γκρέσλε, εδώ υπάρχει περιθώριο για συζήτηση και μάλιστα πολύ υγιή πολιτική συζήτηση. Εάν η Κομισιόν συνεργάζεται με τον ΟΗΕ πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι το κάνει γιατί είναι ο καλύτερος η καλύτερη δυνατή επιλογή αυτή. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο ερώτημα. Το monitoring για τα προγράμματα βοηθείας που διαχειριζόμαστε μέσω του ΟΗΕ. Δεν είναι επαρκές. Δεν είναι επαρκές, διότι η Γούδου, η και η EuroPaid δεν ταυτίζονται. Βέβαια, το πρώτο θέμα που πρέπει να εξετάσει η Κομισιόν είναι να εξετάσει πυλώνα-πυλώνα σύμφωνα με το δημοσιονομικό κανονισμό. Αυτό το έκανε, το κάνει, εξετάζει ακριβώς ποιοι θα γίνουν οι έλεγχοι και οι προμήθειες και και αυτό το έκανε και μετά κάνει δικό της monitoring ε, παίρνει τις εκθέσεις του ΟΗΕ, αλλά τι διαπιστώσαμε εμείς. Διαπιστώσαμε ότι η Κομισιόν δεν έχει ακόμη καταφέρει να έχει επαρκή πληροφόρηση από τις εκθέσεις αυτές του ΟΗΕ. Και τότε τίθεται το ερώτημα. Αν οι εκθέσεις αυτές του ΟΗΕ συμπληρώνονται από πληροφορίες της ίδιας της Κομισιόν, αυτές οι πρόσθετες πληροφορίες είναι και αυτές επαρκείς. Ούτε αυτές. Ούτε αυτές είναι επαρκείς. Οι εκθέσεις του ΟΗΕ γενικά μπορούμε να πούμε ότι είναι υπερβολικά γενικές, δεν αναφέρουν τα προβλήματα που συνάντησαν, συχνά είναι, δημοσιεύονται καθυστερημένα και δεν μας λένε τι πέτυχαν τα σχέδια και τα προγράμματα. Υπάρχει λοιπόν περιθώριο για πολύ σοβαρή κριτική εδώ. Και τώρα δύο λόγια για την Επιτροπή Εξωτερικών Ελεγκτών που όπως όλοι γνωρίζετε έχει αμφισβητήσει το δικαίωμα της Κομισιόν να χορηγήσει πάνη. Η Κομισιόν απ' την άλλη λέει ότι οι δικοί της έλεγχοι αρκούν. Αλλά η Επιτροπή αυτή δεν πήρε από την Κομισιόν επαρκή πληροφόρηση που να το αποδεικνύει αυτό. Ως ελεγκτικό συνέδριο μπορώ να σας πω ότι και εμείς συναντήσαμε δυσκολίες για τη χορήγηση πληροφοριών από τον ΟΗΕ και από τις οργανώσεις του. Τα προβλήματα λοιπόν, για να το πω έτσι, συνεχίζονται. Υπάρχει περιθώριο και για ακόμη περισσότερη συζήτηση εδώ. Τέλος, θα στραφώ σε ορισμένες συστάσεις μας τι συστήνει το συνέδριο στο κεφάλαιο 4 της έκθεσής μας. Λέμε ότι η Κομισιόν πρέπει να δημοσιεύσει συνοπτικές κατευθυντήριες γραμμές όπως τα πρακτικά κριτήρια που ανέφερα προηγουμένως είναι πιο απλή έκφραση αυτή για τη λήψη των αποφάσεων της δεύτερων για το monitoring να ζητήσει εκθέσεις από τον ΟΗΕ που να δείχνουν ποια είναι οι επιπτώσεις των προγραμμάτων και τα αποτελέσματά τους. Κατ' εμάς η Κομισιόν θα έπρεπε επίσης να συνεχίσει να ψάχνει μία διαβεβαίωση, έναν τρόπο να διασφαλίζεται ότι τα προβλήματα πληροφόρησης θα λυθούν. Αυτό είναι το κύριο θέμα που τίθεται ακόμη και ίσως να οφείλεται στην οτροπία ή την ατμόσφαιρα που επικρατεί στις οργανώσεις του ΟΗΕ που τόσο μας αρέσουν. Ίσως να υπάρχει πρόβλημα στάσης εκεί και να τραπείας. Τέλος, το συνέδριο ζήτησε από την Κομισιόν να βρει και άλλους τρόπους συνεργασίας με τον ΟΗΕ για να είναι πιο αποτελεσματική. Τώρα επανέρχομαι σε αυτά που είχε πει η κυρία Γκρέσλε. Η Ένωση η Κομισιόν θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον ΟΗΕ και πώς, αν ναι πώς. Πιστεύω ότι στην έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, άμα τη διαβάσετε προσεκτικά, δεν θα βρείτε μεν τα ονόματα όλων των οργανισμών και οργανώσεων του ΟΗΕ, αλλά άμα το διαβάσετε προσεκτικά θα καταλάβετε ότι παρά το ότι όπως είπα και στην αρχή μπορεί να τα λέμε και καλυμμένα ότι επικρίνουμε πάρα πολύ τον τρόπο συνεργασίας της Ένωσης με τον ΟΗΕ και τα ποσά που δαπανήθηκαν για αυτό το σκοπό που διπλασιάστηκαν πρόσφατα νομίζουμε ότι δεν δικαιολογούνται. Πρέπει λοιπόν να το ξαναδούμε αλλά και στο Κοινοβούλιο και στην Κομισιόν μάλλον παρά στο ελεγκτικό συνέδριο. Εμείς τα είπαμε. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Πρόεδρε, έχοντας ακούσει όσα μα είχε, είχε να μας πει ε, η, το Ελληνικό Συνέδριο, θα ήταν καλύτερα να ακούσουμε πρώτα την Κομισιόν και μετά μας. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Η Κομισιόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φαίνεται ότι οι ε, συναντήσεις με το Ηνωμένο Εθνή οκληρώνονται με το να θαυμάζουν οι μεν τις εκθέσεις των ΔΕ. Αλλά από την άλλη μεριά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε αυτή την έκθεση του ηλεκτρικού Συνεδρίου του 2009 και τον τρόπο με τον οποίο η κυρία Γκρέσλι αντιμετώπισε το θέμα ξεκάθαρα. Τα θέματα που έχουν θυγεί όμως είναι πάρα πολύ σημαντικά και οδήγησαν σε άμεση δράση. Εμείς δεν περιμέναμε να λάβει η χώρα αυτή η συνάντηση για να δράσουμε και θα επανέλθω. Καταρχήν να σας εξηγήσω σε ποιο περιβάλλον εργαζόμαστε. Δηλαδή έχουμε δύο πολιτικά και γραφειοκρατικά σύνολα που το καθένα λειτουργεί ε, με το δικό του τρόπο. Έχουν την πραγματικότητα της Νέας Υόρκης και την πραγματικότητα των Βρυξελών. Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω ούτε τους μένα ούτε τους δε. Αλλά καμιά φορά υπάρχει, ε, υπάρχει πρόβλημα με τη στάση τον μεν και Εδώ πέρα λένε ορισμένοι μην έχετε εμπιστοσύνη απλώς στο ΝΟΙΕ, να πάτε στην Νέα Υόρκη και να δείτε πώς λειτουργεί. Το ίδιο ισχύει με τις Βρυξέλλες. Στη Νέα Υόρκη λένε μην αποδώσετε ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την έκθεση. Εμείς έχουμε ένα σύστημα λογαριασμών, το δικό μας σύστημα και δεν πρόκειται να ακολουθήσουμε αυτά που λένε οι άλλοι. Είναι δύσκολη κατάσταση στα πλαίσια τα οποία είμαστε αναγκασμένοι να εργαστούμε. Δεν πρέπει να συμμορφώσουμε δύο ομάδες κανόνων και η πραγματικότητα των Βρυξελών δεν είναι κάτι που μπορεί να επιβάλλουμε στη Νέα Υόρκη. Δική τους πραγματικότητα έχουν εκεί που θα πρέπει οπωσδήποτε κάπως να λειτουργήσει. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να αναζητήσουμε εταιρικέ σχέσεις σε επίπεδο ενωμένων Εθνών. Παραδείγματος, χάρη αυτά τα ταμεία που δημιουργούνται και πάλι το θέμα είναι ότι εμείς δεν ορίζουμε τίποτα σε επίπεδο ε, εργασίας αλλά οργανώνεται από τους υψηλά ειστάμενους. Υπάρχει ένα πρόβλημα κάπου στον κόσμο, είναι ας έχουμε ένα ε, πρόγραμμα, ένα ταμείο με πολλούς δωρητές και ας προχωρήσουμε. Στο θέμα του μέσου επιστημιστικής βοήθειας, αυτό το κοινοβούλιο μας έδωσε αρκετά στοιχεία στα χέρια μας για να μπορέσουμε να επιμείνουμε προς το ΝΟΙΕ και να του ζητήσουμε να μας κάνει μια ανάλυση χώρα προς χώρα όσον αφορά την ασφάλεια της τροφοδότησης με τρόφιμα. Και επίσης μπορούσε έτσι και το ΙΕ να εφαρμόσει την πολιτική του των Ενωμένων Ενωμένων Εθνών, μπορώ να το πω έτσι. Υπάρχουν βέβαια και καταστάσεις κατά τι οποίε η παραδοσιακή συνεργασία που έχουμε διακόπτεται για λόγω κάποια κρίση. το ότι γίνεται μετά από διαμάχες το θέμα της ουδετερότητας των Ηνωμένων Εθνών είναι επίσης στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη και να μας κάνουν να συνεργαστούμε μαζί τους. Ε, και συνεργαζόμενοι μπορούμε να συμβάλλουμε σε μεγάλες πρωτοβουλίες και όσον αφορά το δημοσιονομικό τομέα και όσον αφορά τις δομές διακυβέρνησης. Αυτό είναι σημαντικό για τη θέση της Ευρώπης και την ορατότητα της Ευρώπης. Ε, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα και συνεχή προβλήματα συνεργασία με το Ηνωμένα Έθνη. Αλλά από τότε που συνεργαζόμαστε εδώ και τέσσερα χρόνια μπορέσαμε να βελτιώσουμε και από τις δύο πλευρές. Έχουμε πάνω της μία συνάντησης ανά για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε τις ε, ατζέντε μας και να έχουμε κοινά αποτελέσματα. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Το θέμα της αναμετρότητας. <coughs> Έχουμε ε, κάποιες κατευθυντήριες γραμμές που εφαρμόζουμε. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες οδηγίες πώς θα φροντίσουμε ώστε όλοι να ξέρουν τα χρήματα που παίρνουν είναι χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm. Είναι πιο αυστηροί σήμερα οι κανόνες για τη βελτίωση των ε, λογιστικών ελέγχων από τα Ηνωμένα Έθνη και θα το ξαναεξτάσουμε με τα Ηνωμένα Έθνη φέτος όσον αφορά τις γραμμές για τους ελέγχους αυτούς. Πριν προωθήσουμε χρήματα σε οποιαδήποτε διεθνή οργάνωση, εξετάζουμε τις διαδικασίες για τον δημοσιονομικό έλεγχο. οι κανόνες εφαρμόζονται αυστηρά, οι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν ε, μα αρκεί να τους επιβάλλουμε στην αρχή, αλλά ελέγχουμε κατά διαστήματα. Έχουμε το δικαίωμα να ελέγχουμε και επιτόπου ότι τα χρήματα που δίνονται έχουν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες και τον Απρίλιο του 2009 συμφωνήσαμε στους ε, κανόνες αναφοράς για, την, ε, για τον έλεγχο. Καμιά φορά υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβαση. Αυτό είναι πολύ ατυχέ. Και το έχουμε ξανασυζητήσει με του αρμοδίου των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά όπω κάθε πολύπλοκο σύστημα υπάρχουν ε, κανόνες γενικού ελέγχου που καμιά φορά βέβαια οι κανόνες αυτοί απλώς μπαίνουν σε ένα ε, φάκελο και δεν τι διαβάζει κανένα. εάν το Ελεκτρικό συνέδριο μας πει ότι είναι σημαντικό αυτό, ε, τότε προσπαθούμε κάτι να κάνουμε στη Νέα Υόρκη και πετυχαίνουμε να έχουμε πρόσβαση σε μερικές ώρες. Δεν είναι ιδανική η μέθοδος αυτή. Όπως είπε και ο κ. Σπίξτερ από το Ελεκτρικό συνέδριο, στο παρελθόν τα επιχειρήματα για τη συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη δεν ήταν ρητά αναφερμένα στην προετοιμασία συμμετοχή σε κάποιο σχέδιο. Το 2008, από το 2008 είπαμε ότι δεν θα υπάρχει πια συζήτηση για κανένα ε, οικονομικό σχέδιο, για καμία χρηματοδότηση, εάν δεν έχουμε αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την συνεργασία στην περίπτωση αυτή. Οι Ηνωμένα Έθνη ανέλαβαν την ε, φετινή ετήσια συνεδρίαση την ε, υποχρέωση να μας ε, δίνουν τα στοιχεία που χρειάζομαστε. Είναι δύσκολο αυτό, αλλά μας δώσουν αυτή την διαβεβαίωση. Περιμένουμε να μας δώσουν τα πρώτα στοιχεία, γιατί αυτή η συμφωνία μόλις επιτεύχει τον Ιούνιο. Μετά περάσαμε αμέσως στις θερινές διακοπές και περιμένουμε τώρα να συνεχίσουμε. Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες ΠΟΠΤΙΑΣ ε, θέλουμε να εξετάζουμε τα αποτελέσματα να είμαστε σίγουροι ότι τα χρήματά μας χρησιμοποιούνται σωστά και αποδίδουν μια αξία. Παραδείγμα χάρη όσον αφορά τα, τα, τα χρήματα που δίνονται για το Ιράκ και το Αφγανιστάν που έχουν στοιχεία που είναι ε, δημόσια προσβάσιμα. Ξέρουμε λοιπόν ότι είναι σημαντικό και για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο να ξέρει σε όλες τις τι γίνεται και να μπορέσει να βελτιώσει το πολιτικό περιβάλλον και το γραφειοκρατικό περιβάλλον. Δεν μπορούμε βέβαια εξ αυτών να προχωρήσουμε γλίγορα, αλλά κάνουμε μικρά για κάθε χρόνο. <laughs> Τέλος για το θα πρέπει πραγματικά να αναγνωρίσουμε ότι στην προκειμένη περίπτωση ήταν πάρα πολύ πολύπλοκο το ε, θέμα και ήταν δύσκολο να δούμε ποιος ήταν υπεύθυνο λόγω των, της μεταφοράς των νομοδοτήτων ε, εξαιτίας των, ε, ε, των αλλαγών που έλαβαν χώρα στις οργανώσεις που εκάστοτε ήταν επιτόπου αρμόδιες. γιατί όλα γινόταν τότε με ταχύτητα και υποπίεση. Η ερευνητική ομάδα που εγκαθιδρύθηκε το 2003 από την ταερωμένη την Όλαφ και τη Μονάδα ε, Οικονομικών Ελέγχων ήταν υπεύθυνη για τον έλεγχο παρατυπιών που αφορούσε κυρίως ε, την ε, κατασκευή στην Πριστίνα. Στο τέλος, το 2008, όλες οι υποθέσεις είτε είχαν κλείσει ή είχαν παραμείνει ακόμα κρεμείς μεταφέρθηκαν στην μονάδα ULEX τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το φορόν η Κομισιόν θέλησε να ρωτήσει τι έγινε όσον αφορά τι δύο περιπτώσει με τις μέβασε σε Άμεν. Η Κομισιόν παραμένει σε στενή συνεργασία και με τα δύο αυτά όργανα, η e ULEX επιβεβαίωσε ότι όλες οι περιπτώσεις που έκλεισαν έχουν περάσει τώρα στα αρχεία από τις ε, ε, αρχές του Κωσυφοπεδίου και δεν υπήρχε τίποτα εκκρεμές όταν μεταφέρθηκαν οι φάκελοι αυτοί από το ΑΜΕΚ στο EULEX. Αυτή τη στιγμή, με την εμπλοκή των Ηνωμένων σε αιτήσια προγράμματα, ε, είναι μονάχα ως συμβαλόμενο μέρος σε μικρά ε, σχέδια. Και η αρμοδιότητα του ελέγχου παραμένει στα χέρια της Κομισιόν. Ελπίζω να σας έδωξα ε, απαντήσεις σε όλα τα θέματα που θίξατε. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ. Η κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ. Είναι βεβαίως Παρακαλώ, μιλάει κανεί με την Κομισιόν. Τώρα θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για το κοσμοπέδιο. Το τελευταίο μου γραπτό ερώτημα για πληροφορίε δείχνει πράγματι πω απασχολείται εδώ πέρα η Λέξα. αλλά από ό,τι μου λέτε μπήκε στο, μπήκαν περιπτώσεις στο αρχείο και έχουν κλείσει. Εντάξει, είναι καλό να καρτάει κανείς αρχείο, αλλά βλέπετε εδώ πέρα πως το μυστικό της επιτυχίας είναι η επανυποβολή. Δηλαδή θα ήθελα να γνωρίζω για αυτές τις περιπτώσεις που επεξεργάστηκε η ITF δεν μπορούμε πλέον να ελπίζουμε τίποτα, δεν θα συμβεί και τίποτα. Έτσι καλά να σας κατάλαβα. Ευχαριστώ, Γκέιρ. Να είμαι λίγο αγενής γιατί νομίζω πως ε, Λείπει η φωνή μου από την Επιτροπή Προϋπολογισμού, αλλά νομίζω πως... Λείπει η ψήφος μου, συγχωρείτε, από την Επιτροπή. Λοιπόν, Εάν μου επιτρέπετε να συνοψίσω, συμφωνείτε σε μεγάλο βαθμό με την εκτίμηση του ελεγκτικού συνεδρίου, επισημαίνεται πως η Νέα Υόρκη, αν θέλετε, είναι ένας άλλος κόσμος που έχει δικούς της νόμους και πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη, αλλά συμφωνείτε με τους φόβους ε, και τις παρατηρήσεις της κυρίας Γκρέσλε με εξαίρεση φόβο αναγνωρίζω πράγματι πως σε πάρα πολλά σημεία στα οποία ε, ασκώ ε, έχετε κάνει πρόοδους και, ε, αν κατάλαβα καλά, στο σημείο που λέμε πως πρέπει να διασφαλίσουμε πως τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου όταν μιλάμε για διάθεση μέσω των υπηρεσιών του ΟΗΕ πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη λογοδοσία. Εκεί πέρα συμφωνούμε. Και αν κατάλαβα καλά, θα ήθελα να μου πείτε... που θα δούμε την ε, καλή διάθεση του ΟΗΕ για να μας βοηθήσει, αν θέλετε, γιατί θα μπορούσαν παραδείγματος χάρη να συνδέσουμε την καταβολή ορισμένων ποσών με κάποιες ε, παραχωρήσεις, δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να συμβιβάσουμε και να έρθει πιο κοντά ο κόσμος αυτός που είπατε της Νέας Υόρκης στον κόσμο των Βρυξελών. Αυτά θα ήθελα από εσάς, δηλαδή να μας πείτε που θα μπορούσαμε να κατευθύνουμε αυτά τα κονδύλια για να μπορέσει και η γραφειοκρατία του ΙΕ να ανταποκριθεί κάπω στι δικέ μα απαιτήσει. Σα ευχαριστώ. Τον λόγο έχει η Κομισιόν για να κλείσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το οποίο είπε η κυρία Γκρίσλε και το πώ αντιλαμβάνεται την κατάσταση σε σχέση με την ίδια λέξη είναι σωστή. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Οπωσδήποτε θα ακολουθήσουμε τις ε, παρατηρήσεις του κύριου Γκάιερ και στη Νέα Υόρκη αυτά τα πράγματα είναι μοιρασμένα στον προπολογισμό. Δεν είναι ένα μέρος που είναι οι συνεισφορές στο σύστημα του ΟΗΕ. Είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης πολλών ανθρώπων σε πολλές περιπτώσεις, αλλά εμείς έχουμε τη γενική εποπτεία στη EuroPaid και θα φροντίσουμε τις ανησυχίες αυτές να τις μεταφέρουμε στον ΟΗΕ. Αυτά μπορώ να πω. Ευχαριστώ. Καλώς τελειώσαμε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και περνάμε τώρα στο τελευταίο σημείο. Έχουμε μία ακρόαση με θέμα την πρόταση οδηγία για την ποινική προστασία οικονομικών σφαιρότων που είναι μπλοκαρισμένα στο Συμβούλιο. Deutsch,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 Θα αρχίσουμε με την ακρόαση που γνωρίζετε. Να μην σας τα ξαναλέω. Πρώτα θα κάνουμε μία συνοψούλα των θεμάτων που εκκρεμούν ακόμη μεταξύ της Επιτροπής μας και της Επιτροπής ε, του Προϋπολογισμού, ιδιαίτερα για την ποινική προστασία. Των οικονομικών συμφερόντων τη κοινότητα και πρόταση κανονισμού για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων τη κοινότητα. Για όσου δεν το ήξεραν γιατί είναι προφανές ότι εδώ θέλουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στη χρησιμοποίηση των δημοσίων πόρων και την καταπολέμηση των απατών, των ατασταλιών, των παρατυπιών, όλα αυτά να διευθετηθούν νομικά. Για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε, κάνουμε και πρόληψη των απατών και να υπάρξει άριστη, βέλτιστη χρησιμοποίηση των δημοσίων πόρων. Άρα πρέπει να υπάρξει κάποιος κανονισμός, οδηγία, κάτι τέλος πάντων και να υπάρχει και ένα ποινικό πλαίσιο επαρκές κυρώσεις. Και όλα αυτά για να μπορέσει επαρκώς να υπάρξει καταπολέμηση της διαφθοράς και της απάτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι και δικό μας θέμα αυτό της Επιτροπής μας, δεν είναι μόνο του εισηγητού. Διότι η αποτελεσματική καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος είναι μία από τις προϋποθέσεις για την καλή χρησιμοποίηση των κοινοτικών ταμείων. Δυστυχώς το Συμβούλιο συνεχίζει να καθυστερεί και να μας θέτει προσκόμματα εμείς όμως πρέπει να επαναλάβουμε την πολιτική μας θέληση να προοδεύσουμε επ' αυτού και να αποδειχθούμε πρωτοπόροι. Η πολιτική θέληση των χωρών μελών επίσης δεν είναι βέλτιστη ορισμένων ιδίως για την καταπολέμηση των απατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ είναι κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον πολίτη και την πολίτησα. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω τον σημερινό μας εισηγητή, τους σημερινούς μας εισηγητές, τον κύριο Λόταρ Κούλ, που είναι υπεύθυνο της Γενικής Διεύθυνσης για το σχεδιασμό στην Όλαφ και έναν εκπρόσωπο από ένα πανεπιστήμιο της Ουγγαρίας και κάποια άλλη κυρία από το Πανεπιστήμιο της Κατάνης. Για μας η ακρόση αυτή θα είναι πολύ χρήσιμη. Υπάρχει λοιπόν εδώ παρόν ο εισηγητής κύριος Ντόιτς που θα είναι και ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι κυρίες και κύριοι. Στόχος ε, της ακρόασης αυτής είναι να επιτευχθεί κάποια πρόοδος σε σχέση με τις ε, προτάσεις που στόχο έχουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών αλλά κολλάνε έξι χρόνια η μία και εννέα χρόνια η άλλη για να μπουν στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου. Είναι λοιπόν προς το κοινό μας συμφέρον να προστατεύεται η κοινότητα από τη διαφθορά, την απάτη και το ξέπλυμα χρημάτων που πλήττουν τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Η απόφαση 2001 κάθος 01 κάθος 05 ε, αφορά τις περιπτώσεις που δεκαλύπτονται από το άρθρο 325 της συνθήκης θα ορίσει τις αξιόπινες πράξεις, τις ποινές και το ποιοι θα διωχθούν και θα έστειν ένα συμβούλιο για το πώς ε, θα γινόταν ο χειρισμός αυτών των υποθέσεων. Ο δε φάκελο 2001 2001-02 αφορούσε την ε, διοικητική αρρωγή μεταξύ των ε, κρατών μελών και θα έδινε μια επιπλέον αρμοδιότητα σε αυτούς φορείς κατά πολέμησης της απάτης αλλά καμία εξουσία έρευνας στην Κομισιόν ή στον Όλαφ. Πρόκειται αυστηρά περί αλληλοβοήθειας διοικητικής. Γιατί βεβαίω αντιλαμβάνεστε πω έχει καταστεί πιο δύσκολη η ανείχνευση των εγκλημάτων αυτών. Ελπίζω λοιπόν με αυτή την ακρόαση να δοθεί νέα ορμή στην διαδικασία. Ω εισηγητή καταβάλω κάθε προσπάθεια να προωθήσω αυτή την διαδικασία και ελπίζω πως η Επιτροπή μας θα μπορέσει να εκφράσει μια κοινή πολιτική βούληση και να ενισχύσει αυτή τη διαδικασία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εδώ πέρα ολοκληρώνω την παρέμβασή μου για να ξεκινήσει η ακρόαση. Ευχαριστώ κύριε Ντόιτς. Τον λόγο στον κύριο Σαουντάσκας, επικεφαλής του γραφείου του κυρίου Σεμέτα που είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο και την καταπολέμηση της απάτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση αυτή για να μιλήσω στην Επιτροπή σας. Ο κύριος Σεμέτα, ο Επίτροπος, Δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει δύο φορές σήμερα στην Επιτροπή σας, ειδικά τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι πολίτες απεργούν, ε, εξασκούν τα δικαιώματά τους και τα αεροδρόμια έχουν κλείσει. Οπότε είναι, ήταν δύσκολο να παραβρεθεί. Η προστασία βεβαίως ε, των οικονομικών συμφέροντων της κοινότητας είναι κεφαλαίου σημασία και είναι θετικό που έχουμε αυτή την ακρόαση για να συζητήσουμε το τι θα γίνει τώρα που έχουμε μια νέα νομική βάση πρέπει να συζητήσουμε λοιπόν αυτές τις δύο προτάσεις. Ε, πρώτα απ' όλα θα δούμε την οδηγία για την ποινική προστασία και μετά για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή. Όσον αφορά λοιπόν την οδηγία για την ποινική προστασία, είναι λυπηρό το ότι η διαδικασία κύρωσης αυτού του μέσου του τρίτου πυλώνα περί προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της κοινότητας χρειάστηκε τόσο χρόνο έτσι ώστε δεν μπόρεσε να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στην προτινόμενη οδηγία αφού υιοθετεί και η έκθεση του Κοινοβουλίου. Να επισημάνω όμως πως η Κομισιόν ήταν συνεπής από όταν παρουσίασε την πρόταση του 2002. Δύο εκθέσεις αξιολόγησης για την εφαρμογή της σύμβασης από τα κράτη-μέλη και πρωτόκολλα στο Εθνικό ε, Ποινικό Δίκαιο ευθύθηκαν το 2004 και 2008 και ήδη έχει αποσταλεί σειρά επιστολών στα κράτη-μέλη εκείνα στα οποία η Κομισιόν θεώρησε πως έπρεπε να γίνει για να ζητήσουμε περαιτέρω πληροφορίες. ή εκθέσεις ε, βρήκαν κάποιες ελλείψεις στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκαν τα πρωτόκολλα από κάποια κράτη-μέλη. Μιλάμε για την εφαρμογή, τον ορισμό της απάτης, ε, των ποινικών κυρώσεων και την ποινικοποίηση, την ποινικοποίηση της διαφθοράς. Ε, η Κομισιόν δεν έλαβε όλες τις απαντήσεις τις οποίες ε, ζήτησε, οπότε μπορεί να χρειάζεται περαιτέρω δράση. Και ενώ η διαδικασία κύρωσης του παλαιού μέσου του τρίτου πυλώνα έχει προχωρήσει, η Τσεχία και η Μάλτα ακόμα δεν έχουν κυρώσει, κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο έξι χρόνια μετά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα λοιπόν έχουμε μία νέα στιβαρή βάση σύμφωνα με την νέα συνθήκη και το άρθρο 235 που έχει διαφορετική διατύπωση από το παλαιό άρθρο 280. Το 280 επέτρεπε για μέτρα στην ε, πρόληψη και την καταπολέμηση τη βλάβη των οικονομικών συμφερόντων τη ε, κοινότητα για να προστατευτούν αυτά στα κράτη-μέλη, αλλά τα μέτρα αυτά δεν αφορούσαν ε, την εφαρμογή του εθνικού ποινικού δικαίου ούτε την ε, εθνική λειτουργία της δικαιοσύνη, ένας περιορισμός ο οποίος έχει αρθεί πλέον στο άρθρο 325. Ο Επίτροπος, ο κύριος Μέτα, οπωσδήποτε θα ήθελε να ακούσει σήμερα τους ε, κυρίους και τις κυρίες βουλευτές για να δει πώς θα μπορέσει να προωθήσει αυτόν τον νομοθετικό φάκελο στο μέλλον και οπωσδήποτε δεν θεωρεί πως μπορούμε απλά να αποσύρουμε την πρόταση. Κατά την άποψή του η πρόταση θα πρέπει είτε να επικαιροποιηθεί είτε να αντικατασταθεί μια πρωτοβουλία που θα βασίζεται στο άρθρο 325 ζήτησε από τις υπηρεσίες του μαζί με τις υπηρεσίες της Αντιπροέδρου Ρέντινγκ να δουν εάν είναι απαραίτητη αναθεώρηση της ε, πρώτας οδηγίας και ενημέρωσή της. Με τη βοήθεια του Κοινοβουλίου ο Επιτροπός είναι επιπισμένος πως θα μπορέσουμε να επιτύχουμε πρόοδο και στο Συμβούλιο. Τώρα, να αναφερθώ στη δεύτερη πρόταση για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή. Πρώτα απ' όλα να υπενθυμίσω την τρέχουσα κατάσταση για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή στην προστασία των οικονομικών σφαίρων της κοινότητας. Και γιατί καλωσορίζουμε αυτή την ακρόαση αφενός, η Κομισιόν το 2004 ξεκίνησε αυτή την πρόταση ενό σχετικού κανονισμού που στόχο έχει δημιουργία ενό γενικού πλαισίου για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων προβλέπει πως τα κράτη-μέλη και οι κομισιόν θα συνεργάζονται, θα συντονίζονται, θα αλληλοβοηθούνται και θα ανταλλάσσουν πληροφορίες σε οτιδήποτε αφορά απάτη εις κοινότητα χωρί. Ε, χωρίς ε, ε, ανεξαρτήτως βεβαίως της λυπής νομοθεσίας και του κανονισμού 515 του 2007. Οπότε θα έχουμε απάτες και στον τομέα των ε, εσόδων και των δαπανών, του ΦΠΑ, διακοινωτικές απάτες, ε, καθώς επίσης ε, και την πρόταση αναδιατύπωσης νομοθεσίας και ζητήματα που σχετίζονται με το πλήσιμο χρημάτων. Από την άλλη, όπως ξέρετε, τον Ιούνιο στο Συμβούλιο τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε ένα πολιτικό συμβασμό για τον κανονισμό 1798 του 2008 για τον τομέα του ΦΠΑ που προβλέπει συνεργασία των αρμοδίων αρχών στην καταπολέμηση της απάτης ΦΠΑ επιπλέον για να προωθηθεί η πολυμερή συνεργασία συστήνεται η Eurofisk, ένα δίκτυο εθνικών υπαλλήλων, οπότε τώρα θα πρέπει να προωθηθεί η αμοιβαία διοικητική συνδρομή στο πλαίσιο του επαναδιατυπωμένου κανονισμού που συνέστησε τη Eurofisk. Επίσης να αναφέρω τις τρεις επιλογές που έχει μπροστά της Κομισιόν για να δώσει συνέχεια στην πρόταση για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή. Επιλογή υπαριθμών 1 να εγκαταλειφθεί η φιλοδοξία ανταλλαγή πληροφοριών για τον ΦΠΑ και να αποσυρθεί τελείω η πρόταση. Η δεύτερη επιλογή να αντικατασταθεί ή να επικυρωποιηθεί πρόταση κανονισμού από μια νέα πρόταση για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή που θα αποκλείει την απάτη ΦΠΑ από το πεδίο εφαρμογής είτε για ένα περιορισμένο διάστημα τριών ετών μέχρι το να αξιολογηθεί το σύστημα ΦΙΣΚ. Εδώ πέρα προκύπτει το ερώτημα του εάν ο κανονισμός αυτός είναι πραγματικά απαραίτητο στον τομέα του ΦΠΑ, εάν ο ΦΠΑ εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής. Μας είπε ο Όλαφ πως η ανάγκη παρέμβαση στα διαρθρωτικά ταμεία είναι περιορισμένη, καθώς περισσότερες περιπτώσεις είναι εθνικές και δεν απαιτούν ε, συνεργασία. Οπότε η περίπτωση των διαρθρωτικών ταμείων θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στον 515 τον αναδιατυπωμένο για την ε, αρρωγή στα, στο του και τον γεωργικό και η τρίτη επιλογή είναι να αναβληθεί τελείως μια απόφαση. Μετά τη συμφωνία λοιπόν για τον κανονισμό. Ίσως φαίνεται πρόωρο να λάβουμε απόφαση για τον νέο κανονισμό που θα συμπεριλαμβάνει τον ΦΠΑ όσον αφορά το ΦΠΑ. Πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση που θα αναλύει το κόστος και το όφελος της ε, ανάμειξης της Κομισιόν σε στρατηγικές αυτές ε, αποφάσεις που θα απαιτήσει οπωσδήποτε πρόσθετους πόρους. Αυτό σημαίνει πως θα λάβουν υπόψη τα μαθήματα που έχουν αντληθεί από την μέχρι τώρα αμοιβαία διοικητική συνδρομή και συνεργασία και το τι πρέπει να κάνει η ομάδα Eurofisco όταν θα αρχίσει να λειτουργεί. Η επικαιροποίηση λοιπόν της ε, πρωτοβουλίας 2004-2006 θα έχει τα εξής πλεονεκτήματα. Πρώτον, θα υπερασπίζει συνεπώς ένα υποχρεωτικό σύστημα αμοιβαίας συνδρομής και για απάτη ΦΠΑ και για τα διαρθρωτικά ταμεία μέσω κομισιών και και του Όλαφ βεβαίω, σύμφωνα με το άρθρο 305 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επιβάλλει νέες υποχρεώσεις αναφορά στα κράτη-μέλη πέραν από την ανταλλαγή πληροφοριών για τις λεγόμενες μεγάλες υποθέσεις και οπωσδήποτε δεν θα επηρεάσει το πεδίο εφαρμογή του αναδιατυπωμένου οργανισμού. Δεύτερον, θα έχει μια ευρύ, ένα ευρύτερο πεδίο εφαρμογή σε αντίθεση με τον κανονισμό που καλύπτει μόνο τον ΦΠΑ. Θα καλύπτει όμω μόνο τι περιπτώσει μεγάλη απάτη που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την Ένωση. Και τρίτον, θα δώσει ένα πιο προληπτικό ρόλο στην Κομισιόν, η οποία θα διευκολύνει τα κράτη-μέλη μέσω μιας πλατφόρμας, αλλά θα συμμετέχει πλήρως και στην ανταλλαγή πληροφοριών. Σύμφωνα λοιπόν με τον ε, αναδιατυπωμένο κανονισμό, η ανταλλαγή πληροφοριών θα οργανώνεται από τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν θα παρέχει μόνο διοικητική υποστήριξη αλλά όχι επιχειρησιακή. Όπως βλέπετε λοιπόν κυρίες και κύριοι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις μας. Αναμένουμε λοιπόν τις θέσεις σας και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και αν έχετε άλλες ερωτήσεις είμαι σίγουρος πως ο συνάδελφός μου θα μπορέσει να σας απαντήσει. Και γρατσίε μόλτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σαντάουσκας. Θα δώσουμε τώρα τον λόγο στον κύριο Κιούλκ, επικεφαλής της ε, Μονάδας Γενικής Πολιτικής του Όλαφ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω έτσι λίγες ε, παρατηρήσεις και εγώ για να συμπληρώσω αυτά τα οποία ακούστηκαν. Νομίζω είπε αρκετά πράγματα ο επικεφαλής του γραφείου του κυρίου Σεμέτα. Απλά θα ήθελα να πω πως πρέπει να είναι σωστό το ότι βλέπουμε αυτές τις δύο προτάσεις μαζί στην ημερήσια διάταξη γιατί πράγματι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε συνολικά και αφορά το πλαίσιο λειτουργίας του όλα. Και εδώ πέρα είναι δύο ζητήματα αυτά που ήταν πάντα ευαίσθητα στο παρελθόν. Δηλαδή αφενός το θέμα του μέχρι σε ποιο βαθμό μπορεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να περιέχει ποινικά θέματα και δεύτερον τι μπορεί να γίνει στον τομέα της απάτης του ΦΠΑ και ποια είναι η εντολή της Κομισιόν στον τομέα αυτών με βάση την ε, συνθήκη για την καταπολέμηση της απάτης πιο ειδικά. Τώρα για την προστασία των οικονομικών σφαίρων της κοινότητας βλέπω τρεις προκλήσεις. Εάν δούμε το τι θα πρέπει να γίνει από εδώ και μπρος. Μιλάμε για ζητήματα ουσιαστικού ποινικού δικαίου αλλά και ζητήματα συνεργασίας μεταξύ Όλαφ και των αρχών δίωξης και έρευνας και μια άλλη προπτική, μια προπτική θεσμική, δηλαδή η προετοιμασία της εφαρμογής μιας διάταξης στη συνθήκη που αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κάποιες παρατηρήσεις λοιπόν σε αυτές τις ε, προκλήσεις που νομίζω πρέπει να τις δούμε μαζί. Πρώτα απ' όλα το πώς θα συγκλίνει το δίκαιο στον τομέα του ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Ο κ. Σαντάσκας είπε πως εδώ πέρα έχουμε ήδη νομικά μέσα του τρίτου πυλώνα τα οποία μετά από επίπονες ε, διαδικασίες κύρωσης ετέθησαν στην αρχή αυτής της δεκαετίας του 2002 επιτέλους εν ισχύ και έχουμε και το δεύτερο επιπρόσθετο πρωτόκολλο με την κύρωση από την Ιταλία το 2008 οπότε βρισκόμαστε τώρα στην φάση, στη διαδικασία της εφαρμογής η Κομισιόν έγραψε δύο ευρύτατες εκτεταμένες εκθέσεις εν μέρη καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως έχουμε κάποια πρόοδο, αλλά και στο ότι δεν είναι πλήρως ικανοποιητική η κατάσταση. Υπάρχουν προβλήματα ελλείψης ισοδυναμίας και ελλείψης εφαρμογής σε κάποια κράτη-μέλη και συγκεκριμένα δεν έχουμε σε όλα τα κράτη-μέλη το ίδιο αξιόπινο αντικείμενο, αλλά οδηγούμαστε στο να βασιζόμαστε στο ποινικό δίκαιο της ε, κάθε χώρας, κάτι το οποίο βεβαίως μας οδηγεί στο ότι αν έχουμε μια διασυνοριακή απάτη πρέπει να δούμε ποια ακριβώς είναι η αξιόπινη πράξη στη χώρα Χ και στην άλλη οπότε θα πρέπει να δούμε το πώς θα υπάρχει κοινή εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη. Επιπλέον διαπιστώνουμε πως έχουμε μια διαδικασία η οποία θα απασχολήσει την Κομισιόν και το Συμβούλιο και οπωσδήποτε στο προσεχές μέλλον, στο άμεσο μέλλον, για τα κράτη-μέλη εκείνα στα οποία έχει απευθυνθεί η Κομισιόν με επιστολές και λέει πρέπει να μας εξηγήσετε τι έχετε κάνει εκεί πέρα και τι θεωρείτε εσείς ότι είναι οι υποχρεώσεις που έχετε σύμφωνα με την συμφωνία. Αυτό μπορεί να καταλήξει και ενώπιον του δικαστηρίου. Εν πάση περιπτώσει η διαδικασία θα προχωρήσει. Αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι πως και από νομοθετική σκοπιά υπό το φως της θέσης ενισχύς της συνθήκης της Λισαβόνας έχουμε ένα δίκαιο το οποίο θα πρέπει να δημιουργηθεί και να ισχύει άμεσα για να μην περάσουμε ξανά από τη διαδικασία κύρωσης στο κάθε κράτος μέλος. Και αυτή είναι σημαντική πτυχή. Δεύτερον, το δικονομικό δίκαιο. Το άρθρο 325 ανοίγει νέες προοπτικές. Είχαμε την πρόταση της Κομισιόν το 2001 και τότε είχαμε διαχωρίσει το τι μπορεί να γίνει σύμφωνα με το άρθρο 280 που προέβλεπε την εξαίρεση ότι δηλαδή αυτά τα μέτρα δεν μπορούν να αφορούν εφαρμογή του ποινικού δικαίου στα κράτη-μέλη. Οπότε σε μεγάλο βαθμό βαφήσαμε εκτός της ε, περιπτώσεις συνεργασίας από το κεκτημένο του τρίτου πυλώνα. Οπότε θα πρέπει να δούμε ποια είναι η συνεργασία μεταξύ όλαφ και διοκτικών αρχών σε μια μελλοντική πρόταση και τι μπορούμε να κάνουμε και με την μεταρρύθμιση του Όλαφ. Με βάση το άρθρο 325, από ό,τι φαίνεται μπορούμε να πάμε τουλάχιστον πιο μακριά από ό,τι μέχρι στιγμής και τρίτον και σύντομα. Εάν έχουμε εδώ πέρα την προοπτική μιας μελλοντικής ε, ε, διοκτικής και ερευνητικής αρχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει το ζήτημα του ποιο θα πρέπει να είναι το νομοθετικό πλαίσιο αυτής της αρχής, ποιες θα είναι συγκεκριμένα οι αρμοδιότητες τους, οι ουσιαστικές. Γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα μέσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο το οποίο θα μας λέει για ποιες ποινικέ διαδικασίες είναι αρμόδιος ο Ευρωπαίος εισαγγελέα, για ποια δικήματα υπό ποιες συνθήκες και θα πρέπει να προετοιμαστούμε γιατί μία μέρα θα το συναντήσουμε αυτό ως πρόκληση στο νομοθετικό πεδίο και βεβαίως αυτή είναι μια κάπως ε, μια προοπτική που θα τη δούμε περισσότερο στο μέλλον αλλά στο άρθρο 3.25 θα πρέπει νομίζω πάντα αυτό να το ερμηνεύουμε σε συνδυασμό με το άρθρο 86 τη συνθήκη. Όσον αφορά τώρα τον ΦΠΑ και το σχετικό κανονισμό και την αμοιβαία συνδρομή. Και εδώ πέρα βλέπω τρεις προκλήσεις. Η πρώτη πρόκληση είναι να ξεκαθαρίσει το νομικό πλαίσιο, το οποίο εξακολουθεί ε, δυστυχώς να είναι αντικείμενο διαμάχης με το Συμβούλιο. Δεύτερη πρόκληση, η επιχειρησιακές ανάγκες σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν και η τρίτη πρόκληση είναι αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Σαντάουσκας να σκεφτούμε μια ε, να δούμε δηλαδή ποια θα είναι η νομοθετική ευκαιρία που θα δούμε πρώτα απ' όλα το νομικό πλαίσιο ο λόγος για τον οποίο είχαμε τόσο μεγάλες δυσκολίες εκ των προτέρων στο Συμβούλιο για να σημειώσουμε κάποια πρόοδο για να αποδεχτούν τα κράτη-μέλη πως θα πρέπει να υπάρχει εδώ πέρα μια Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασίας των οικονομικών συμφερόντων η οποία θα δραστηριοποιείται στον τομέα του ΦΠΑ βασίζεται βεβαίως τους ε, περιορισμούς του ορισμού των ε, ατασταλιών οι οποίες βεβαίως αφορούν μόνο τους παραδοσιακούς ίδιους πόρους. Βεβαίως όσο εξελίσσεται το νομικό πλαίσιο προστασίας των οικονομικών σφαιρών υπάρχει ένας διχασμός μεταξύ των πραγμάτων που πέφτουν εντός του ορισμού των ανομαλιών αυτών και καλύπτονται από τον Όλαφ και του τομέα του ΦΠΑ που δεν συμπεριλαμβάνεται στους παραδοσιακούς ίδιους πόρους σύμφωνα με τον ορισμό αυτών. Ταυτόχρονα όμως είναι σαφές πως και το 209α της συνθήκης του Μαστρίχτ και το 288 ή το 325 σύμφωνα με τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας ερμηνεύονται ως εξής τα οικονομικά συμφέροντα αφορούν πρώτα απ' όλα όλων τον προϋπολογισμό, όλες τις δαπάνες, αλλά βεβαίως και όλο το πεδίο εφαρμογής των ίδιων πόρων. Και σύμφωνα με την, ε, τις αποφάσεις του 10 αφορούν γενικά τα συμφέροντα της κοινότητας. Οπότε έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι κάποιο στρεβλή, δηλαδή το τι όρισε ως νομοθέτη, ο νομοθέτης ως προστασία των οικονομικών συμφέροντων της κοινότητας και καταλήξαμε με το ΟΕΡΟΦΙΣΚ και τον κανονισμό των επαναδιατυπωμένων να προσεγγίσουμε και να συγκλίνουν οι διατάξεις στον τομέα των φορολογικό. Βεβαίως αυτό δεν μας αρκεί γιατί μιλάμε, πως, ε, μιλάμε βεβαίως για συμφέροντα κοινά των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα γιατί αν θέλει να συνεργαστεί με τις φορολογικές αρχές των κρατών μελών ο Λαφή όταν του ζητάνε να συνεργαστεί το πρώτο ερώτημα που τίθεται είναι με ποια νομική βάση. Και το μόνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι πως υπάρχει ένα άρθρο 325 που καλύπτει γενικώ τα οικονομικά συμφέροντα και τα οικονομικά συμφέροντα συμπεριλαμβάνουν και τον ΦΠΑ. Και υπάρχει λοιπόν μια γενική εντολή για να συνεργαστεί η Κομισιόν με τα κράτη-μέλη, αλλά βεβαίως αυτό δεν φτάνει πάρα πολύ για να δικαιολογήσει συγκεκριμένη ροή πληροφοριών. Οπότε αυτές είναι οι προκλήσεις και δεν μπορούμε βεβαίως να ξεπεράσουμε αυτή την ασάφεια και να πούμε πως η Κομισιόν έχει εδώ πέρα μία εντολή να λειτουργεί επιχειρησιακά με τα κράτη-μέλη. Δεύτερον, βεβαίως είναι η αναγκαιότητα δράσης και αυτό βεβαίως ήταν και αντικείμενο ακρόασης στην Επιτροπή σας το 2008 που επιβεβαιώθηκε και από τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια στις εκθέσεις τους πως απαιτείται στον τομέα της απάτης ΦΠΑ να υπάρχει ένα, μια υπηρεσία clearing σε ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία θα μπορέσει να προσφέρει την δυνατότητα συνεργασίας στα κράτη-μέλη εκεί όπου είναι υποχρεωμένα να το κάνουν αυτό και συνολικά να προσφέρει την δυνατότητα πολύπλευρης ανταλλαγής ε, πληροφοριών. Παραδείγματο χάρη όταν μιλάμε για την απάτη καρουσέλ, δυστυχώς δεν το καταφέραμε αυτό και βεβαίως τώρα υπάρχει το ερώτημα, εξακολουθεί να υπάρχει μία ανάγκη δράσης ε, τη στιγμή στην οποία το Συμβούλιο ομολογουμένως μετά από δύσκολες διαπραγματεύσεις ε, κατέληξε στο Eurofisk και στην νέα οδηγία και ενώ ξέρουμε πως για τα κράτη-μέλη είναι κόκκινο πανί να υπάρχει επιχειρησιακή ανταλλαγή πληροφοριών με την Ταξιούδη, την Κομισιόν. Και είναι βεβαίως πολύ πολιτικό το ζήτημα. Θεωρώ πως θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα αυτό κάνοντας χρήση του κανονισμού Eurofisk που νομίζω είναι προς εφαρμογή, είναι αύριο νομίζω στην ε, ημερήσια διάταξη της Κορεπέρ. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα τοποθετηθούν τα κράτη-μέλη, θα υπάρξουν διάφορες ομάδες εργασίας. Μετά υπάρχει το Eurocanet, ε, κομισιόν με τη συμμετοχή του Βελγίου και θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό και βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο επίσης δεν πρέπει να παραμελήσουμε και αφορά το ζήτημα των προτεραιοτήτων του Όλαφ. Γνωρίζουμε πως σε πάρα πολλούς τομείς υπάρχουν προτεραιότητες, γνωρίζουμε πως έχουμε κάποιες και πρέπει να δράσουμε, ακόμα και αν επικεντρωθούμε μόνο σε μεγάλες περιπτώσεις, οι οποίες χωρίς μια επένδυση ποσών και προσωπικού δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν. Οπότε είναι ζήτημα βεβαίως ε, και της κατάλληλης στιγμής, της χρονικής. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα λάβετε υπόψη και εδώ πέρα θα την τελειώσω την παρέμβασή μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Αρχίζει η συζήτηση για αυτά τα θέματα. Φαντάζομαι οι συνάδελφοι θα θέλουν να θέσουν ορισμένα ερωτήματα ή απορίες. Ο αντιπρόεδρος Στάις πρέπει να φύγει, γι' αυτό ίσως η συζήτηση να καθυστερήσει και να ακούσουμε πρώτα όλες τις εισηγήσεις ο καθηγητής Κάς στο Ίδρυμα Ποινικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Μίσκο στην Ουγγαρία. Ευχαριστώ. Παρακαλώ συγχωρήστε με που θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα αλλά τι να κάνω, μου είναι πιο εύκολο. Εγώ είμαι εμπειρογνώμων στο ποινικό δίκαιο. Εδώ και 13 χρόνια και είμαι μέλος μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης Προστασία των συμφερόντων τη Ένωση με όμως και καθηγητής ποινικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Μίσκο. Νομίζω ότι οι ριζικές αλλαγές, οι ριζικότερες αλλαγές που σημειώθηκαν τελευταία ήταν αυτές που προέβλεψε η συνθήκη της Λισαβόνος. Εκεί τι είδαμε, είδαμε μια σειρά μια σειρά προσπαθειών, διαπραγματεύσεων και ορισμένων συμβιβασμών που βρίσκονται στην πρόταση οδηγίας ήδη από το 2001. Έχουν αλλάξει τα πράγματα βέβαια και είμαι βέβαιος ότι τώρα αντιμετωπίζουμε μία μοναδική ευκαιρία μια μοναδική ευκαιρία μία μοναδική ευκαιρία γιατί άλλαξε η νομοθεσία και τα πρότυπα. Και τα πρότυπα. Και τα πρότυπα όσον αφορά ιδιαίτερα την προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Εγώ δεν έκανα καμία διαβούλευση προηγουμένως με τον κύριο Κουλ, αλλά ένα από τα μηνύματα που θέλω να σας δώσω είναι το εξής που συμφωνεί και με εκείνον. Τώρα που η συνθήκη της Λισαβόνας έχει καταργήσει τη δομή σε και η νέα αρχή είναι η αμοιβαία αναγνώριση που θεωρείται και θεμελιώδης αρχή από τη συνθήκη αυτήν. Ας πούμε στο 325, στο άρθρο 325 που καταργεί την παράγραφο 4 του προηγουμένου άρθρου 280, που έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επηρεάσει το εθνικά δικαστικά συστήματα και τον ποινικό τους κώδικα. Όλα αυτά έχουν αλλάξει. Η πρόταση οδηγίας του 2001 που βασιζόταν, βασιζόταν σε ένα συμβιβασμό. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ίδια η νομοθεσία δημιουργεί ευκαιρίες ή και δεσμεύσεις, υποχρεώσεις για ένα κράτος μέλος ώστε αυτό να ξέρει ξέρει ότι οποιαδήποτε παραβίαση των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ένωσης θα τιμωρείται αυστηρά. Επίσης ισχύει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να κάνουν πολλά για αυτό το θέμα, πάρα πολλά. Ξέρουμε ότι τα εθνικά ποινικά δίκαια, οι κώδικες ποινικού δικαίου, που είναι ένα από τα τελευταία προπύργια της εθνικής κυριαρχίας θεωρούνται από τα κράτη ως ποκόριο φθαλμού. Η διαφορά των ποινικών δικαίων των χωρών μελών είναι όμως ένα από τα εμπόδια για την επίτευξη για την επίτευξη του στόχου της εναρμόνισης της νομοθεσίας και των διαδικασιών. Αν και σε προηγούμενες φάσεις δεν υπήρξε καμία πραγματική δυνατότητα ή ευκαιρία να επιδείξει η Ένωση ή κάποιο κράτος περισσότερη ορμή για την εναρμόνιση των ποινικών διώξεων εγκληματιών, ακόμη και αν πρόκειται για την παραβίαση των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, στο τομέα της δικαιοσύνης, οι δυνατότητες της Ένωσης έχουν διευρυνθεί. και πρόκειται για πολύ αποτελεσματικό εργαλείο πρόοδου. Το επόμενο σημείο που θέλω να θίξω αφορά τις διαδικασίες. Χωρίς τους θεσμούς, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, παρά το γεγονός ότι οι ιδιοκτικές αρχές των κρατών ορίζουν πώς και πότε θα δράσουν ή θα αντιδράσουν, Χωρίς λοιπόν αυτά, η συνθήκη της Λισαβόνας ε, μας έχει δημιουργήσει νέες δυνατότητες και ευκαιρίες. Δεν ισχύει πια ούτε ο η τριπυλωνική δομή, ούτε, ούτε τα υπόλοιπα. Και έτσι δίνεται η δυνατότητα στενότερης συνεργασίας. Και τώρα που δεν είναι πια απλώς ιδέα η έννοια του ενωσιακού εισαγγελέα, αλλά μια πραγματική δυνατότητα που δίνει το ενωσιακό δίκαιο, νομίζω ότι δίνεται η δυνατότητα στην Ένωση έτσι να δράσει πιο ενωτικά και στο διαδικαστικό τομέα. Αυτό βέβαια προϋποθέτει συμβιβασμούς. Επειδή δεν είμαι μάντης δεν μπορώ να σας πω ποιες άλλες δυνατότητες μπορεί να ανοίξουν κατά τις διαπραγματεύσεις. Νομίζω όμως ότι είναι ρεαλιστική η πρώτη η πολύπλο το πολύπλοκο αυτό νομοθέτημα α, για τη δημιουργία της έδρας του ενωσιακού εισαγγελέως και από τη μία και η συνεργασία Όλαφ και Eurojust από την άλλη αυξάνεται έτσι γίνεται πιο αποτελεσματική προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Ε, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Grazie. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο καθηγητής από την Κατάνη. Η καθηγήτρια μας συγχωρείτε. Ε, ευχαριστώ. Μια αποσαφήνιση καταρχάς. Δεν έχουμε πολύ χρόνο και γι' αυτό θα επικεντρωθώ στην πρόταση οδηγίας που αφορά την ποινική προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ένωσης. Θα προσπαθήσω την παρέμβασή μου να την δομήσω σε τρία σημεία. Πρώτον, ορισμένα γενικά σχόλια για τις νέες δικαιοδοσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ποινικό τομέα που απορρέουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεύτερον, το νομικό υπόβαθρο μιας πιθανής μελλοντικής οδηγίας που να αφορά την προσέγγιση των ε, εθνικών ποινικών προτύπων για την προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ένωσης και τρίτον οι προοπτικές έγκρισης σύντομα μια τέτοια οδηγία. Ας αρχίσω όμως από την αρχή. Γενικές παρατηρήσεις για τις νέες ποινικέ δικαιοδοσίες της Ένωσης. Γνωρίζουμε τη συνθήκη της Λισαβόνας όπως μας το υποθύμησε και ο καθηγητής Φαρκάς, για πρώτη φορά ρητά ορίζει οι δικαιοδοσίες της Ένωσης σε περιπτώσεις πρωτοβουλειών εναρμόνισης νομοθεσίας, ποινική νομοθεσίας των κρατών μελών. Πρέπει εδώ να αποσαφηνίσω, αλλά το ξέρετε όλοι είμαστε πυρογνώμονες εδώ, ότι καμία διάταξη της συνθήκης της Λισαβόνας δεν δίνει, δεν χορηγεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποινική δικαιοδοσία καθεαυτήν. Καμία ρήτρα της συνθήκης σήμερα δεν επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκρίνει διατάξεις που να έχουν πραγματικό χαρακτήρα ποινικού δικαίου άμεσης εφαρμογής υποχρεωτικά από εθνικούς δικαστάς. Αυτό όμως που προβλέπει είναι κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Το άρθρο 183 για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου φαίνεται ότι η Ένωση μέσω της οδηγίας δηλαδή ενός δεσμευτικού νομοθετήματος προηγουμένως επρόκειται για τον πρώτο πυλώνα τώρα είναι δεσμευτικό νομοθέτημα επιτρέπεται στην Ένωση να εγκρίνει ελάχιστα πρότυπα ποινικών κυρώσεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πρώτον, ορισμένες υποθέσεις τομείς δηλαδή ιδιαίτερους τομείς εγκληματικότητας με διεθνή χαρακτήρα και προβλέπεται ολόκληρος κατάλογος εκεί και δεύτερη σειρά περιπτώσεων που είναι πολύ πιο λεπτά θέματα για τα κράτη-μέλη, δηλαδή όλες τις περιπτώσεις όπου η σύγκληση των εθνικών ποινικών διατάξεων θα ήταν απαραίτητη για να υπάρξει εγγύηση μιας αποτελεσματικότερης αντιεγκληματικής πολιτικής της Ένωσης. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, εφόσον τα κράτη εγκρίνουν την οδηγία, τότε τα κράτη πρέπει να υποβάλουν συγκεκριμένο ορισμό των συμπεριφορών που θέλουν να κυρώσουν και με σεβασμό φυσικά όλων των υπολείπων διατάξεων της οδηγίας. Εάν όμως ο νομοθέτης δεν ακολουθήσει τις υποχρεώσεις ποινικοποίηση της οδηγίας, τότε μπορεί να συρθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Με προσφυγή επί παραλήψη. Βεβαίως. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να έχει τεράστιες επιπτώσεις στις εθνικές συμπεριφορές. Το άρθρο 183 πρέπει να σας το ξαναπώ αφήνει έναν πολιτικό φραγμό προστασίας και διπλωματικό στην παράγραφο 3 του προβλέπει ότι ένα κράτος όταν θέλει να μπλοκάρει μια τέτοια νομοθετική διαδικασία μπορεί να το κάνει εφόσον θεωρηθεί ότι το προτινόμενο πρότυπο μπορεί, μπορεί να θίξει ουσιώδεις πτυχές του δικαστικού συστήματος της χώρας αυτής. Εδώ ανοίγεται ένας πολιτικο-διπλωματικός δρόμος στο Συμβούλιο για να μπορέσει να εφαρμόσει ενισχυμένη συνεργασία. Είναι πάντως προφανές ότι όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα κάνουν από αυτή τη ρήτρα τα κράτη-μέλη. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος ακριβώς η σημασία της δικαιοδοσίας αυτής για την προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ένωσης και περνάω έτσι στο δεύτερο μου σημείο το νομικό υπόβαθρο Μία πιθανή μελλοντική οδηγία όπου είχα αναφέρει προηγουμένως. Λοιπόν, αν παραμείνουμε στο άρθρο 83 λέει τώρα η ομιλήτρια που προβλέπει ρητά αυτήν την περίπτωση την δυνατότητα παρέμβασης στον ποινικό τομέα της Ένωσης τότε η προστασία των δημοσιονομικών συμφωνών δεν καλύπτεται. Δεν καλύπτεται από αυτή τη δικαιοδοσία και θα ήταν τελείως περίεργο κάτι τέτοιο. Γιατί, διότι δεν υπάρχει καμιά αναφορά της απάτης, καμία μνήα της απάτης ή άλλων παρανόμων δραστηριοτήτων ως κάτι που παραβιάζει τα δημοσιονομικά, βλάπτει τα δημοσιονομικά συμφέροντα της Ένωσης και έτσι υπάρχει ο κίνδυνος η παράγραφος 2 του 83 να εφαρμοστεί. Εδώ πρόκειται για πρόβλημα. Και εδώ συμφωνούν μάλλον όλοι. Είναι πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Και ίσως αυτό γίνεται με την παραπομπή στο άρθρο 325 που συνεχίζει το πρώην 180. Το άρθρο αυτό όπως και το 280 λέει τώρα η ομιλήτρια ε, θεωρείται ως ε, εφαρμοστική ρήτρα για την καταπολέμηση του οργανωμένου κλίματος σύμφωνα με ορισμένα συγκεκριμένα κριτήρια που καθορίζουν το κατά πόσο είναι η κοινωτική διαδικασία. Γιατί, διότι μία από τις αντιρρήσεις που ακούμε συχνά ως τη δυνατότητα παρέμβασης της Ένωσης του τομέα αυτών βασίζεται στο ότι η προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων δεν αναφέρεται ρητά στο άρθρο 83 και λένε ότι εδώ πρόκειται για ερμηνεία που μπορεί κανείς να την κάνει και στενά και με στενή ερμηνεία δεν νομιμοποιείται παρέμβαση νομικού τύπου από την Ένωση για πρότυπα που προβλέπουν τέτοια ενωσιακή νομοθεσία. Αφού δεν αναφέρεται λοιπόν η καταπολέμηση της απάτης, Φαίνεται ότι δεν είναι και πολύ εγγυημένη η δυνατότητα αυτή παρέμβαση της Ένωσης. Όταν όμως μιλάμε για μέτρα καταπολέμησης της απάτης συνδεόμενα με την προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της Ένωσης, τότε η οδηγία που προβλέπει η σύγκληση των προτύπων των κρατών μελών σύμφωνα με το 385 325 με συγχωρείτε αυτό θα σήμαινε ότι οτιδήποτε αφορά το ποινικό δίκαιο των χωρών μελών απαγορεύεται από την Ένωση να τύχει παρέμβαση. Σας λέω μόνο τα σημαντικότερα τώρα λοιπόν παρέμβαση με βάση το 325 δεν γίνεται, αλλά από την άλλη μεριά θεωρείται υποχρεωτική. Άρα χρειάζεται εδώ περαιτέρω αποσαφήνιση, γιατί στο 325 δεν γίνεται λόγος για ελάχιστα πρότυπα, ενώ γίνεται στο άλλο. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει εδώ κάποια αποσαφήνιση. Και τρίτο και τελευταίο, ακόμη και σημαντικό, πιο σημαντικό, για να καταλάβουμε μέχρι πού φτάνει η δικαιοδοσία της Ένωσης, το 325 δεν αναφέρει πουθενά τέτοια, ούτε καμία κατεπίουσα διαδικασία. Άρα, ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την εξαίρεση αυτή που είχε προβλεφθεί αρχικά. Άρα η δικαιοδοσία αυτή είναι πολύ πιο προωθημένη και θεμητή με τον έννοια του 325 διότι τα δημοσιονομικά συμφέροντα της Ένωσης από τη φύση του την ίδια είναι διεθνικού χαρακτήρα. Αυτό ως απάντηση το, στις αντιρρήσεις που συχνά ακούω. Είναι λοιπόν δυνατόν να ακουστεί ως αντίρρηση το περιεχόμενο της προτινομένης οδηγίας, διότι δεν πρόκειται μόνο για τη στενή έννοια της απάτης, αλλά και για ανακύκλωση, διαφθορά, δωροδοκία, όπως τα ορίζει το 325-4, το οποίο αναφέρει μόνον πολέμηση και πρόληψη της απάτης. Άρα θα μπορούσε κανείς να πει ότι η αντίρρηση ισχύει και ότι άλλη πρέπει να είναι η νομική βάση το 83 με τα όρια και τους περιορισμούς που έχει αυτό. Εξάλλου, εξάλλου λέγω, ούτε το 325, ούτε το 83, ούτε ο συνδυασμός τους δεν μπορούν να επιτρέψουν την έγκριση σχετικού κανονισμού, δηλαδή πράξεις άμεσα εφαρμοστέας στα κράτη-μέλη. Άρα ένα τέτοιο εργαλείο δεν χρειάζεται. Δεν θα χρειάζεται όταν θα υπάρξει αυτή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τότε όμως θα χρειαστεί αλλαγή των συνθήκων και θα πρέπει να γράφει ρητά ότι υπάρχει αυτή η δικαιοδοσία. Τέλος. Πρέπει, σύντομα βέβαια, σύντομα, να δούμε εάν σήμερα υπάρχουν οι δυνατότητες, οι προϋποθέσεις για να μπορεί να εγκριθεί μια οδηγία που να εισάγει σύγκληση του ποινικού δικαίου των χωρών μελών. Κατ' εμέ, Είτε, προ... είτε μιλήσουμε είτε βασιστούμε στην έννοια του σεβασμού της αρχής της ultima ratio, δηλαδή κάτι που ούτως ή άλλως πρέπει να το αναφέρουμε αν μιλήσουμε για ποινικέ δικαιοδοσίες και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω και αν είναι έμεσες οι, οι δικαιοδοσίες αυτές, αφού πρέπει να περάσουμε από, το εσωτερικό, από την εσωτερική νομοθεσία, πρέπει να γίνει σεβαστή και η αρχή της επικουρικότητας. Τώρα, η ultima ratio. Αφού πρόκειται για δημοσιονομικά συμφέροντα, όλοι καταλαβαίνουν πόσο σημαντικά είναι αυτά αν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβιώσει και να είναι αξιόπιστη, πρέπει να γίνει λόγος για την Ούλτιμα τη Είναι Θα μπορούσε κανείς να πει ότι συμπεριφορές που βλάπτουν το αγαθό αυτό του δημοσιονομικού συμφέροντος πρέπει να τιμωρούνται και μάλιστα υποχρεωτικά διότι αν υπολογίσει κανείς τα υπέρ και τα κατά, διαπιστώνει αμέσως και εύκολα ότι μόνο ποινική μπορεί να είναι η κύρωση αυτή. Αυτό είναι αναπόφευκτο συμπέρασμα. Θυμηθείτε τι είπε προηγουμένως ο Τμαρκούλ, ότι από τις διάφορες αξιολογήσεις που βλέπουμε να έχουν γίνει ως προς την εφαρμογή του πρώην τρίτου πυλώνα φαίνεται ότι όχι απλώς μερικές χώρες δεν έχουν μεταφέρει την νομοθεσία αυτή της δικαιότητα αλλά δεν υπάρχει αρκετή αποτελεσματικότητα και στις χώρες που την έχουν μεταφέρει. Έτσι λοιπόν πρέπει να γίνει μια πραγματική σύγκληση ποινικών προτύπων. Η Κομισιόν μάλιστα λέει ότι ένα από τα ζωτικότερα στοιχεία του ορισμού της ενίας της απάτης είναι κάτι που αφήνει ακόμη να περνάνε τεράστιες διαφορές απαρατήρητες. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν η α ή β συμπεριφορά συμπεριλαμβάνεται στον ορισμό ή όχι. Πιστεύω λοιπόν ότι ακόμα και με βάση την αρχή της επικουρικότητας οι προϋποθέσεις για να μπορεί νομικά μια, η Ένωση να παρέμβει ποινικά υπάρχουν και έτσι θα έχει τη δυνατότητα να είναι πολύ αποτελεσματικότερη. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον φίλο του κ. και να δω αν θα μπορέσει να απαντήσει πώς μπορούμε να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τα δημοσιονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν δεν επιβάλλουμε κυρώσεις ποινικέ και πολιτικές με μέτρα που εγγυούνται την ανωνυμία των οικονομικών συνεργών. Τις έχω κατά νου εδώ κάτι που απέ αποφάσισε η Ιταλική κυβέρνηση ένα μέτρο που δεν επιτρέπει την πληρωμή του ΦΠΑ και επιτρέπει να επανέλθουν με ένα ποσοστό φόρου 5% χρήματα που ήταν σε ε, φορολογικούς παραδείσους και ανώνυμα πάντα. Τι γίνεται λοιπόν σε περίπτωση απάτης. Έθεσα το ερώτημα αυτό πλιστάκι προς την Κομισιόν και θα ήθελα κάποια στιγμή να πάρω μια απάντηση. Δεν βλέπω πως να υπάρχει κανένας εδώ στην Κομισιόν να μου απαντήσει. Σας παρακαλώ να μεταβιβάσετε την ερώτηση με αυτή στον κύριο Σεμέτα και ελπίζω και η Όλαφ να μπορέσει να ασχοληθεί με το θέμα αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και που είναι αντίθετο με την πούληση προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της κοινότητας. Ε, <clears throat> ε, <clears throat> ε, Ευχαριστώ πολύ. Ε, ε, λυπούμε που ο κ. Σαντάσκο σα αναγκάστηκε να φύγει γιατί είχε μια, κάποια άλλη ελμένη υποχρέωση. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί κανένας να δει πόσο σημαντική είναι η συνεργασία στην καταπαλώμηση της απάτης στο φορολογικό τομέα γενικά και ειδικότερα στο τομέα ΦΠΑ. Το πρόβλημα βέβαια δεν έχει επιληθεί. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω και είναι και πολύ επίκαιρο είναι ότι η Κομισιόν τα περασμένα 10 χρόνια περίπου ξεκίνησε να διαπραγματεύεται συμφωνίες συνεργασίας με εκείνες τις τρίτες χώρες οι οποίες είναι γνωστές σαν οικονομική παράδειση και που στο παρελθόν δεν ήταν πολύ συνεργάσιμη. Αυτό το 2004 με μια συμφωνία με την Ελβετία για την καταπολέμηση των απατών. Που η συμφωνία αυτή είναι προσωρινά εφαρμόσιμη, δεν έχει τεθεί σε ισχύ, γιατί είναι μια μεικτή συμφωνία που πρέπει να επικυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη. Από την άλλη μεριά επιτρέπει μια συνεργασία με τις φορολογικές αρχές της Ελβετίας σε όλες τις υποθέσεις ε, απάτης ΦΠΑ και φοροδιαφυγής ε, ΦΠΑ και όσον αφορά επίση απάτε με τους ειδικού φόρους κατανάλωσης. Ξεκινώντας από αυτό έχουμε μια συμφωνία με το Λίχτενστάιν. Και αυτή είναι μια συμφωνία που προχωράει πέρα από τη συμφωνία με την ε, Ελβετία γιατί προβλέπει γενικά τη συνεργασία στον φορολογικό τομέα και προβλέπει έντονες υποχρεώσεις συνεργασίας με το Λίχτενστάιν γενικά όσον αφορά τους υποκείμενους σε φορολογία που συμμετείχαν σε κάποιες επενδύσεις στο Λίχτενστάιν. Το Λίχτενστάιν πρέπει να δίνει τι σχετικές πληροφορίες. Δυστυχώς δεν έχει εξεταστεί αυτό το θέμα που ξεκίνησε από πέρσι που βασίζεται στους κανόνες του ΣΑ για την ε, φορολογική συνεργασία αλλά δεν έχει προωθηθεί από το Συμβούλιο. Και μέχρι στιγμής απέτυχε λόγω της αντίστασης του Λουξεμβούργου. Δεν ασχολήθηκε δηλαδή εξ αυτού το Συμβούλιο. Και έτσι η υπογραφή της συμφωνίας δεν έχει ακόμα εγκριθεί από το Συμβούλιο αυτό. Όταν υπογραφεί αυτή η συμφωνία, έχει η Κομισιόν ήδη υποβάλει συστάσεις για διαπραγματευτικέ αντολέ με άλλε τρίτε χώρε, παραδείγματο χάρη Αντόρα, Μονακό, Σαν Μαρίνο. Και επίση μια περαιτέρω διαπραγματεύση με την Ελβετία, πολύ σημαντικό. και θα μπορούν να γίνουν διαπραγματεύσει και με άλλες ε, τρίτες χώρε. αν υπάρχει κάποιο πρότυπο όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και έτσι θα μπορούσαν να οριστούν πρότυπα που θα οδηγήσουν παγκοσμίω όλα τα τρίτα κράτη που ε, είναι φορολογική παράδειση να αναγνωρίσουν τα πρότυμα αυτά. Αυτός είναι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στις πλαίσια δικασία του G20. Έχετε δίκιο όμως, το πρόβλημα δεν έχει ακόμα επιληφθεί. Πολύ ωραία, κύριε ο πρόεδρος. Θέλει κανένα το λόγο? Θέλετε να ολοκληρώσετε? Köszönöm σα ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητέ για τι πολύ χρήσιμες ιδέες και πολύ αξιόλογες ιδέες που υπέβαλαν και που θα μας κάνουν να μελετήσουμε περαιτέρω το θέμα, να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τους στόχους. Αυτές οι δύο οδηγίε είναι πάρα πολύ σημαντικέ για να προστατευτούν τα ε, οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης. και να προχωρήσουμε στην απόφαση του Συμβουλίου να δοθεί δηλαδή μια ορμή ναι. σε, αυτή την, ε, σε αυτό το φάκελο. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, επισκέπτες, θα ήθελα να σας πω ότι βάσει αυτών που ακούστηκαν μπορούμε να διατυπώσουμε ένα ελάχιστο πρόγραμμα αφενός και να έχουμε και κάποια προοπτική μακροπρόθεσμες ιδέες δηλαδή που απαιτούν πολιτική και επαγγελματική υποστήριξη από τη δική μας Επιτροπή. Όπως είπε ο κ. Σανταούσκας, Ε, λόγω της συνθήκης της Λισαβόνας έχουμε διαφορετική κατάσταση και συνεργασία με την Κομισιόν θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες που μπορούμε να καταστήσουμε πιο επίκαιρες, πιο σύγχρονες αυτές τις δύο οδηγίες, να τις επαναδιατυπώσουμε και να μπορέσουν έτσι οι τροποποιημένες οδηγίες να πάρουν το πράσινο φως στο Συμβούλιο. Όπως τα είπαν οι κύριοι καθηγητές, οι εμπεριλαμβάνομενες στις συμβολές τους, συζητάμε εδώ ένα ευρύτερο πλήρες πρόγραμμα Πιστεύω ότι η συνθήκη της Λισαβόνας άνοιξε ένα παράθυρο ευκαιρίας στην νομοθετική μας εργασία με στόχο την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από το 1995, από τότε που υπογράφει η συνθήκη του Μαστρίχτη, πετύχαμε κάποια πρόοδο. Εκ των υστέρων όμως μπορούμε να πούμε ότι βέβαια πέρασαν υπερβολικά πολλά χρόνια για να έχουμε σχετικά μικρά αποτελέσματα πρόοδου. Μετά τη θέση ισχύ της συνθήκης της έχουμε την ευκαιρία βασιζόμενοι στις νέες αυτές νομοθετικές διατάξεις, να προστατεύσουμε καλύτερα τα οικονομικά μας συμφέροντα και να τροποποιήσουμε τμήματα του ποινικού κώδικα και έτσι να δώσουμε νέα μορφή σε εκείνες ε, τις υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι υπεύθυνε για την εφαρμογή αυτών των νόμων. Παραδείγματο χάνει το θέμα της ε, μεταρρύθμισης Όλαφ συζητιέται ήδη. Θα πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι λύσεις για το ε, έργο του δημοσίου κατήγορου. Και η υπηρεσία αυτή του δημοσίου κατηγορού δημιουργεί ένα πλαίσιο για το πρόγραμμα, το PIF 15, Eh, Μας δίνει τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της ε, τρέχουσας ηττίας του Κοινοβουλίου και της ηττίας της δεύτερης Επιτροπής Μπαρόζο βάσω των διευκολύνσεων της συνθήκης της ε, Λισαβόνας να τροποποιήσουμε και τον ποινικό κώδικα και τις υπηρεσίες που ασχολούνται με την εφαρμογή Ακούσαμε πάρα πολύ χρήσιμα θέματα σήμερα. Μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει πολιτική βούληση στην Επιτροπή. Ο ελάχιστο στόχο θα πρέπει να είναι να οι τρει αυτοί που είναι προκαρισμένοι όποιον του Συμβουλίου τώρα και να εξετάσουμε κατά πόσον και πώς μπορεί η Επιτροπή μας να εμπλακεί ενεργά σε μια μακροπρόθεσμη γενική λύση και για τα θεσμικά όργανα και για τον ποινικό κώδικα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους συζητητές και παρουσιαστές και σας